José Κυρία Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την Εθνική Πλατφόρμα των Θυγωμένων από το νόμο περί Με 2.000 ακίνητα, 6.000 ε, 6-7.000 θυγόμενους πολίτες. Πριν από δύο χρόνια υποβάλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια εκτεταμένη αναφορά και αιτιάσει για καταχρηστική εφαρμογή του νόμου περιακτών και μάλιστα πριν από ένα χρόνο υπευλήθηκε έκθεση Άουκεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το θέμα αυτό. Τα τελευταία διετία είχαμε πολλές εξελίξεις. Η κυβέρνηση αγνοεί, μάλλον αρνείται την ύπαρξη αυτού του ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. θεωρεί ότι είναι ψέμα αυτό το επιχείρημα και επίσης δεν μας ε, δεν επιτρέπει στους να εξετάσουν τα δικόγραφα όλων αυτών των υποθέσεων. Εμείς υποβάλαμε στα πολιτικά κόμματα για μελέτη ένα σχέδιο αναθεώρησης του νόμου περιακτών και με συστάσεις ε, που αντιγράψαμε από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαμε να ομοδοποιήσουμε τις καταχρήσεις του νόμου αυτού σε ορισμένες κατηγορίες. Για παράδειγμα, η αναδρομική ισχύ του νόμου περί ακτών. Έχει κανείς μια νόμιμη ιδιοκτησία εκτός του δημοσίου κτήματος, μετά διευρύνεται ορισμός για τη δημόσια περιουσία, επηρεάζεται από τον νέο ορισμό και χάνεται την ιδιοκτησία σας, την περιουσία σας. Επίσης, δεν δίνονται αποζημιώσεις για τις απαλωτριώσει αυτές, τουλάχιστον δεν γίνονται χρηματικές αποζημιώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις και θεωρητικά δίνεται η διοικητική παραχώρηση. Στην πράξη όμως δεν έχουμε ούτε καν αυτή τη διοικητική παραχώρηση, γιατί η κυβέρνηση χορηγεί αυτές τις παραχωρήσεις γενικά μόνο τα χρειάζεται το οικόπεδο για ένα δημόσιο έργο. Δίνει δηλαδή την παραχώρηση και μετά θεωρητικά, αλλά δεν την ε, εφαρμόζει τις περισσότερες φορές μετέτρεψε αυτή την παραχώρηση που κανονικά θα πρέπει να δίνει μια ασφάλεια, νομική ασφάλεια και μια ηρεμία στους πολίτες. Ουσιαστικά η παραχώρηση αυτή είναι σήμα ανησυχία και έλλειψης ασφάλειας δικαίου. Επίσης κατεδαφίζονται νόμιμα κτίσματα. Στις Βαλεαρίδες για παράδειγμα είχαμε ε, μία κατοικία αποκτήστηκε το 1920, ήταν εγγεγραμμένη στο κτηματολόγιο νόμιμους τίτλους και σήμερα έχει εκδοθεί διάταγμα κατεδάφισης. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον ιδιοκτήτη ως εγκληματία, γιατί εκτός ότι έχει διατάξει την κατεδάφιση της οικία, υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να πληρώσει και τα έξοδα που ανέρχονται σε 3.600 ευρώ. Δηλαδή όχι μόνο κατέστρεψαν τη ζωή αυτού του ανθρώπου, τον υποχρεώνουν να, πληρώσουν, να πληρώσει και τα έξοδα κατεδάφισης, αφήνοντας στον δρόμο τον ίδιο και την οικογένειά του. Η, τα δημόσια έργα όπως ο Μαρίνας η λιμάνια εμποδίζουν τη συντηρήση των ακτών. Άρα προχωρεί η, ε, προχωρεί η θάλασσα προς την ξηρά και το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να προβεί σε νέα οριοθέτηση της δημόσιας περιουσίας, πηγαίνοντας όλο και προς τα μέσα στην ξηρά. Έτσι και άλλοι ιδιοκτήτες χάνουν την ε, περιουσία τους, μερικές φορές και από αμέλεια της κυβέρνησης. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που μετά την οριοθέτηση, τη νέα χωρομέτρηση και μετά την απώλεια των περιουσιών, μετά την απώλεια και όχι πριν, τότε είναι που ε, διατάσσεται η αναγέννηση ε, με έργα της ακτής, αφού έχουν χάσει όμως οι άνθρωποι τις περιουσίες τους. Επίσης, οι διάφορες υποθέσεις ε, οριοθέτησης ε, του δημόσιου κτήματος γίνονται αυθαίρετα, γιατί η χωρομέτρηση γίνεται από την κυβέρνηση τελείως αυθαίρετα, χωρίς τεκμήρια, όπου τους καπνίσει στην ουσία. Και εξαιτία ακριβώς τη έλλειψη αποδείξεων έχουμε πολλέ τέτοιε αυθαίρετε οριοθετήσει και χωρομετρήσει στα Κανάρια νησιά. Αυτή η διαδικασία της οριοθέτηση του δημοσίου κτήματο ε, γίνεται εγκρυπτό και παραβίστο. Δεν ενημερώνεται κανένας. Δεν δίνεται καν η δυνατότητα υπεράσπισης στο θυγόμενο. Για να μην μιλήσουμε για την απώλεια του δικαιώματος κυριότητας. Ορισμένες ε, προτάσεις για έργα της, δημόσια έργα της κυβέρνησης, για παράδειγμα για μία αποβάθρα με τη νέα οροθέτηση αν βρίσκεται ένα κτίσμα στο, στην πορεία αυτής της α, ε, βόλτας της παραλίας ή της αποβάθρας, δεν, δεν ενημερώνεται καν έγκαιρα ο ιδιοκτήτης ή δεν έχει κανένα λόγο στην απόφαση αν θα καταδεφιστεί το κτίσμα του ή όχι. Βρίσκεται πρωτοτελεσμένο γεγονότος. Επίσης, ε, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται πολύ αυστηρά σε μία λωρίδα 100 μέτρων, καταδικάζοντας σε αργό θάνατο πολλούς οικισμούς, πολλές παραδοσιακές ε, οικίες, ιδιαίτερα στα Κανάρια νησιά, αλλά και στη Γαλλικία. Και τέλος, ο νόμος περιακτών δεν χρησιμεύσε τελικά για να α, ε, αναχαιτιστεί η ανεξέλεκτη αστική ανάπτυξη στις παραλίες. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα ε, δόθηκε μια τέτοια άδεια για αστική ανάπτυξη στην Καρταχένα. Ενώ κρίθηκε παράνομη μία αντίστοιχη παραλία στην οποία τα κτίσματα ήταν πολύ παλιά και παραδοσιακά. Οι απαντήσεις της κυβερνήσης ήταν θεωρητικές, γενικές και αόριστες. Θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως παραμύθια για παιδιά. Είναι σαν ανούρισμα τα επιχειρήματα που έδωσε η κυβέρνηση. Είναι σαν την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων τα παραμύθια που μας ξεφούρνησε η Ισπανική κυβέρνηση. Γιατί αυτά που μας είπε η εκπρόσωπη της Ισπανικής κυβέρνησης είναι η θεωρία, το ιδεατό. Η πράξη είναι αυτή που σας εξήγησα εγώ. Γιατί δεν θα ερχόμασταν αν δεν είχαμε λόγο στην Επιτροπή σας να ταξιδεύουμε άγρια χαράματα για να σας παρουσιάζουμε την υπόθεσή μας. Αυτή δυστυχώς είναι η σκληρή πραγματικότητα που σας παρουσίασα εγώ. Θα πρέπει να επέμβετε όχι μόνο για να αποκατασταθούν τα δικαιώματα των ε, πολιτών που έχουν παραβιαστεί, αλλά και η ποδοπατημένη τους αξιοπρέπεια ορισμένων πολιτών που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το δικαίωμα ε, να ζει κανείς μέσα στην ευρωπαϊκή επικράτεια τους εξασφαλίζει μια ελευθερία και ασφάλεια. Ευχαριστώ. Grazie. Carmen la Hernandez. Carmen Hernandez. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Κάρμεν Ντελάμο Ερνάντε και εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση των Θυγωμένων από το νόμο τη Ακτή. Είχα ετοιμάσει μία ομιλία για να σα εξηγήσω τι ε, συνθήκε ε, για, το, για, μία συνοικία στον Αλικάντε. Μετά τη χθεσινή παρουσίαση του, της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Κυβέρνησης έχω τροποποίησει την ομιλία μου καταδεικνύοντα τι τεσταλίες τη ισπανική κυβέρνηση. Λάθος μας είπε η εκπρόσωπος τη ισπανική κυβέρνηση ότι οι οριοθετήσει μπορούν να, τύχουν, να, να προσβληθούν με προσφυγή. Λάθος. Ε, επιτρέπεται ε, μόνο στην Αουδιένσια Νασιονάλ τέτοια προσφυγή κατά των αριοθετήσεων. Και μάλιστα το δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει σε δεύτερο βαθμό αυτές τις προσφυγές. Οπότε είναι τελείως ανεδαφικές οι παρατηρήσεις της Ισπανικής κυβέρνησης για το δημόσιο κτήμα. Επίσης, ε, έχουμε το δημόσιο κτήμα στις ε, λωρίδες των ακτών που βρέχονται από τη θάλασσα. Ενώ είναι δηλαδή ο Αιγαίολος ενώ ο νόμος περί ακτών υιοθετεί ένα πολύ αυθαίρετο ορισμό οποιαδήποτε ζώνη θεωρήσει ελκυστική η Ισπανική κυβέρνηση μπορεί να τη χαρακτηρίσει δημόσιο κτήμα. Πολύ αυθαίρετα. Νομίζω ότι αν ήθελε η Ισπανική κυβέρνηση να, να προσπίσει τις ακτές θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να στερεί από τους πολίτες τις νομίμως κτηθήσεις περιουσίες τους. Είναι πολύ αυθαίρετη η εφαρμογή του νόμου αυτού από την Ισπανική κυβέρνηση με ολέθριες συνέπειες για το περιβάλλον. Γιατί παρόλα αυτά, παρά το νόμο αυτό, γίνεται τελείω ανεξέλεγκτη αστική ανάπτυξη σε πάρα πολλέ παραλίε και ακτέ. Άλλωστε, κανεί δεν μπορεί να στερηθεί την περιουσία του χωρί δίκαιη αποζημίωση. Μία παραχώρηση όμως 30 κονταετή δεν συνιστά δίκαιη αποζημίωση. Μοιάζει περισσότερο με δίμευση. Η Ισπανική κυβέρνηση δεν σέβεται την ατομική ιδιοκτησία, γιατί χθε αρνήθηκε το χαρακτηρισμό τη ω θεμελιώδου δικαιώματο. Διαβάστε, κυρία Μαρτίνε, το άρθρο 17 τη Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που λέει ότι κάθε άνθρωπο έχει δικαίωμα στην ατομική και συλλογική ιδιοκτησία και κανεί δεν θα στερηθεί αυθαίρετα τη ιδιοκτησία του. Ακούσαμε χθε επανειλημμένω στην αίθουσα αυτή ότι είναι καλό ο νόμο περί αλλά η η αφαίρετη εφαρμογή του οδηγεί στην ε, παράλογη κατάσταση. Δεν συμφωνούμε όμως, γιατί ένας νόμος που επιτρέπει μία ελαττωματική και ακατάλληλη εφαρμογή και παραβιάζει ε, ευθέω τα δικαιώματα των πολιτών είναι ένας διστραμμένος νόμος και αυτό ισχύει για τον νόμο περιακτών της Ισπανίας. Ο νόμος περιακτών της Ισπανίας ουσιαστικά συνιστά ένα κοινωνικό σκάνδαλο. Θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομεριακά όλες οι αναφορές, όλες οι αιτιάσεις και απευθύνουμε έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει την Ισπανική κυβέρνηση να μην εφαρμόσει τον νόμο περί ακτών που αντιβαίνει στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Οι πολίτες που έχουν θυγεί από τον νόμο αυτό και εμφανίζονται στην Επιτροπή σας είναι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό προσβλέπουμε στην ε, υποστήριξη και συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην προστασία του. Ευχαριστώ. Yeah. με Λέγομαι Κάριν Κόμπερλινγκ, είμαι Γερμανίδα. Ο άντρας μου είναι Βρετανός. Βρίσκομαι εδώ για να σας ε, αναφερθώ ε, στην για να αναφερθώ στην κατάσταση του Πουερτίτο. Το Πουερτίτο είναι ένα ψαροχώρι, ε, βρίσκεται μακριά από άλλες ε, περιοχές. Το 78, 10 χρόνια πριν ε, εφαρμοστεί ε, ο, κόσμος, ο νόμος περί ε, Αιγιαλού, αγόρασα το σπίτι μου το οποίο χτίστηκε τη δεκαετία του 30. δεν είχε σχεδόν δρόμο, δεν είχε νερό, δεν είχε ηλεκτρικό και βρισκόταν μακριά από το λεγόμενο ντομίνιο πουμπλικό. Το 2005 η γραμμή αυτή να διαβάσετε σας παρακαλώ λίγο πιο αργά για τους διερμηνείς. Ωραία. Η διαγράμμιση αυτή άλλαξε το 2005 και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό έγινε χωρίς ε, επίσημη κοινοποίηση ή διαβούλευση των ε, αρμόδιων αρχών και μάλιστα έγινε κατάλογος και μάλιστα ε, εισήχθη άλλο όνομα για την δική μου ε, ιδιοκτησία και έτσι δεν μπορούσα πια να υπερασπιστώ την περιουσία μου. Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό. Οι αρχές είχαν τον αριθμό κτηματολογίου μου, εγώ είμαι η μόνη, από το 1978 ήμουν, ήμουν η μόνη ξένη ε, στο χωριό, ε, όλοι με ήξεραν. Έτσι λοιπόν ε, απαλωτριώθηκε η περιουσία μου και τώρα απειλούν με κατηδάφιση. Μιλάμε εδώ για κατάφορη κατάχρηση των δικαιωμάτων, ιδιαίτερα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Και επίσης βλέπουμε αυθαίρετη και αναδρομική ισχύ του νόμου, εφαρμογή του νόμου η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ε, δώσει άμεσα την παραχώρηση, αλλά αυτό δεν έχει γίνει. Βρίσκομαι σε καθεστώς ε, νομικής απεβαιότητας, δεν έχω ιδιοκτησία, δεν έχω παραχώρηση και δεν ξέρω ποια είναι τα δικαιώματά μου. Ούτε η Ισπανική κυβέρνηση δεν το ξέρει αυτό, διότι ε, η κατάσταση αυτή ρυθμίζεται μέρη από τον νόμο. Ε, μπορεί να μου δοθεί η παραχώρηση αλλά και να μου αφαιρεθεί αμέσως ε, διότι ε, προβλέπεται ένας πεζόδρομος 200 μέτρων σε ένα φυσικό πάρκο και το... Από το Υπουργείο ζητήθηκε άρση του δομήνιο Πούμπλικο και η περιοχή στην οποία προβλέπεται αυτός ο πεζόδρομος θεωρείται παράκτια περιοχή, αλλά ο σχετικός νόμος απαγορεύει τέτοια έργα τόσο κοντά στην ακτή. Για να χτιστεί αυτός ο πεζόδρομος θα πρέπει να μπαζωθεί με τα μπάζα από τα σπίτια που θα κατεδαφιστούν. Ε, μιλάμε για τρομερές ε, περιβαλλοντικές καταχρήσεις. Το παραδοσιακό ψαροχώρι, παρότι δεν ε, είναι η αιτία της καταστροφής, της περιβαλλοντικής καταστροφής, απειλείται. Θα η δημιουργία νέου, ε, νέας διαγράμμισης ε, χωρίς ε, να έχουν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι είναι επίσης μια κατάφορη παραβίαση, όπως επίσης και η παραβίαση των συμβάσεων. Βρισκόμαστε σε νομική αβεβαιότητα. Επίσης το θέμα των παραχωρήσεων είναι παράνομο και η αρχές ε, σε συνεργασία με τις ε, επιχειρήσεις ε, οικοδόμησης εφαρμόζουν αυθαίρετα τον νόμο περί γυαλού και προβλέπουν δημιουργία κάμπινγκ για 375 άτομα, ε, προβλέπουν δημιουργία πεζόδρομου πάνω στην ακτή και ε, άλλα έργα. Υπάρχουν ε, πολλές νομικές αβεβαιότητες εδώ πέρα. Θα ήθελα όμως να πω ότι εδώ και πέντε χρόνια εγώ και η οικογένειά μου νιώθουμε ότι μας βασανίζουμε. Ε, ότι μας βασανίζουν. Ε, αυτό επηρεάζει την υγεία μας, ε, την ευημερία μας και την οικονομία μας. Κάθε μέρα κάνω έρευνες σχετικά με τα αν μήπως απειλείται το σπίτι μου. Αυτό συνεπάγεται σημαντικό κόστος, πόσο μάλλον που όλη η διαδικασία πραγματοποιείται σε άλλη γλώσσα από τη δική μου. Η απειλή είναι τεράστια ε, γραπτός όμως δεν έχω λάβει τίποτα σχετικά με το τι γίνεται. Ε, βρίσκομαι σε ένα τρομερό καθεστώς αβεβαιότητας ε, και απειλούμε. Μιλάμε για διοικητική τρομοκρατία και δεν θα το ευχόμουν αυτό σε κανέναν. Το πορτίτο χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται προσπάθειες για περιβαλλοντική ανάπτυξη που θα λάβει υπόψη το φυσικό πάρκο στην Χαντία. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία ε, με τους ε, κατοίκους. Ε, υποφέρω μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους, Ισπανούς και Ευρωπαίους πολίτες και ελπίζω ότι θα αναγνωριστούν τα δικαιώματα όλων, διότι αυτά είναι τα πρότυπα τα οποία είναι περήφανη η Ευρώπη που έχει θέσει. Ευχαριστώ. Ingeborg Χόφμαν, καλημέρα. Σας ευχαριστώ που ε, ε, που μας ακούτε. Η Αμπούρια Μπράβα ε, βρίσκεται κοντά στην Μπράβα και είναι μια πόλη σαν τη Βενετία. Περίπου 5.000 άνθρωποι επηρεάζονται από την κατάσταση. Πρόκειται για μια ειδική περίπτωση. Δεν μιλάμε για καταστροφή των ακτών ούτε μιλάμε για περιβαλλοντική προστασία. Η Αμπούρια Μπράβα δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 60. Η ακτή έχει ε, πλάτος 500 με 700 μέτρα και πίσω από αυτό βρίσκεται ε, η πόλη μέχρι 3 χιλιόμετρα μέσα στο, ε, στη στεριά. 30 χιλιόμετρα κανάλια υπάρχουν εδώ πέρα όπου μπορεί κανείς να μεταφερθεί με ε, βάρκες. Και ε, προβλέπεται απαλωτρίωση για τέσσερα είδη ιδιοκτησία, ε, κάποια, κάποια ιδιωτικά ακίνητα. λάβανε άδεια ώστε να δημιουργηθούν ιδιωτικοί λιμένες και έχουν εισαχθεί στο κτηματολόγιο. Δεύτερον, ε, υπάρχουν κάποια σπίτια ε, όπου υπάρχουν ε, χώροι για βάρκες. Μιλάμε, για παράδειγμα, για 10 μέτρα οικόπεδο κοντά στη θάλασσα, σπίτι και 8 μέτρα όπου δεν είναι οι βάρκες. Επίσης, υπάρχουν κάποια μέρη όπου ε, ε, ε, έχει δημιουργηθεί χώρος να αφήνουν τις βάρκες μέσα στο οικόπεδό τους και όπου έχουν δημιουργηθεί, σαν να λέμε, γκαράζια τις βάρκες. Θα πρέπει όμως το κτηματολόγιο να διορθωθεί, διότι μιλάμε για απαλωτρίωση, αποζημίωση με παραχώρηση. Δεν είναι το ίδιο ε, με ιδιοκτησία και μας ε, δημιουργεί άλλα προβλήματα η κατάσταση αυτή, στα οποία θα επανέλθω. Το κτηματολόγιο είναι ε, ένα δημόσιο μέσο και είναι η μόνη κρατική εγγύηση για την ιδιοκτησία. Επιστεύτηκαμε το κράτος, πιστέψαμε το κράτος και εμπιστευτήκαμε το κτηματολόγιο. Πιστεύουμε ότι παραβιάζονται τα βασικά μας δικαιώματα. Όταν λάβει κανείς ε, παραχώρηση, ε, δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Τα κανάλια αυτά θεωρούνται ακτή και ε, οι ακτές θα πρέπει να είναι ελεύθερες για το κοινό. Όλα τα... Σε, όλα τα, σε όλες τις ιδιωτικές ιδιοκτησίες θα πρέπει να δημιουργείται πρόσβαση στο κοινό. Αυτό όμως θα αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ε, ιδιοκτησίας ε, των ιδιωτών ε, και θα κατέστρεφε και τους πολύ όμορφους χώρους αυτούς κοντά στην ακτή και επίσης θα καταργηθεί έτσι το δικαίωμά μας για ιδιωτική ζωή. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να καταδαφιστούν αυτοί οι χώροι. επανειλημμένα έχουν αγοραστεί, μεταβιβαστεί ή κληρονομηθεί τέτοια ακίνητα και έχουν εισαχθεί στο κτηματολόγιο χωρίς δουλείες. Όλοι αγόρασαν καλή την πίστη. Εγώ το 1978 αγόρασα την ιδιοκτησία μου στο Ισπανικό προξενείο της Φραγκφούρτης. Το κράτος μέχρι σήμερα ε, εισπράττει φόρους ε, για ε, τις ιδιοκτησίες αυτές. Για παράδειγμα, φόρο κληρονομιάς, φόρο κοινοτικό, φόρο αγοράς ιδιοκτησίας κλπ. Πώς είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνθήκες ιδιοκτησίας να αλλάζουν με τέτοιο θεμελιώδη τρόπο και να εφαρμόζονται ε, οι νόμοι αναδρομικά. Ο ε, νόμος ε, περί Αιγιαλού τέθηκε σε ισχύ το 1988, τότε υπήρχε η Αμπούρια Μπράβα ήδη επί 20 χρόνια και δεν αναγνωρίστηκε κανένα δικαίωμα χρησικτησίας. Το επιχείρημα ότι ο νόμος αυτός του 88 ε, βασιζόταν σε προηγούμενους νόμους, για παράδειγμα τον Λέιντε Άγουας του 1868, δεν αποτελεί ε, δικαιολογία διότι το, κράτος, ε, το ίδιο το κράτος μέχρι το 2008 δεν εφήρμοσε τον νόμο αυτό στην Απούρια Μπράβα. Το κράτος με την εισαγωγή στο κτηματολόγιο νομιμοποίησε επανειλημμένα τις πωλήσει και εισέπρατε σχετικούς φόρους. Η οι ιδιοκτήτε ε, ε, νιώθουν ότι έχουν εξαπατηθεί. Μέχρι το φθινόπωρο του 2008 κανένας ιδιοκτήτη, ε, κανένας συμβολιογράφος, κανένα, κανένα προξενείο και ειδικά όχι το κτηματολόγιο δεν ήξερε τι γίνεται με τις ιδιοκτησίες αυτές. Φοβούμαστε το, στις 29 το του 2088 το Υπουργείο των ε, Ακτών ε, άλλαξε την ε, διαγράμμιση των ακτών και αυτή τη στιγμή το μόνο που απομένει είναι η προσφυγή. Είναι το μόνο μέσο που απομένει. Απαιτούμε να μην εφαρμοστεί ο νόμος περί αγιαλού στην Φιουδάδενα Ναβεγάμπλε Αμπούρια Μπράβα. Θέλουμε προστασία το να εξαιρέσουμε την αμπούρια μπράβα από τον νόμο περί είναι δυνατόν, διότι είναι η μόνη Ciudad Navegable που, ε, έχει δημιουργηθεί, που είναι ε, κατά 100% τεχνητή. Η εφαρμογή του νόμου περί στην αμπούρια μπράβα δεν έχει κανένα νόημα και δεν ε, χρησιμεύει σε κανέναν και δεν ακολουθεί το πνεύμα του νόμου, δεν μιλάμε για προστασία των ακτών, προστασία του περιβάλλοντος ή το δημόσιο συμφέρον. Η μη εφαρμογή του νόμου θα ε, απέτρεπε τόση ζημιά, θα έσωζε τόσες, ε, τόσες ε, περιουσίες. Πολλοί ιδιοκτήτες θέλουν να πουλήσουν, αλλά ποιος θα θέλει να αγοράσει και με ποια εγγύηση. Τη στιγμή που το κτηματολόγιο και το δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν ισχύουν. Σας ζητούμε βοήθεια ώστε να προστατεύσετε τα δικαιώματα ε, ιδιοκτησίας ε, των ε, ιδιοκτητών της Αμπούρια Μπράβα. Θέλουμε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, προστασία του καταναλωτή και σεβασμό του δικαιώματος για ιδιωτική ζωή και ιδιοκτησία. Ευχαριστώ. Grazie. La Ley de Costas veut rendre aux citoyens l'usage des plages et enlever... Ε, ε, ορίζει ότι πρέπει να κατεδαφιστούν ό,τι έχει ε, χτιστεί σε δημόσιο χώρο. Εμάς όμως δεν έχει χτιστεί σε δημόσιο χώρο. Πρόκειται για μια μεγάλο αγρόκτημα με βοσκή στο εσωτερικό της γης. Οι οδοί κατασκευάστηκαν και κανάλια χαράχτηκαν προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στα σπίτια μέχρι 4 χιλιόμετρα στο εσωτερικό. Οι ιδιοκτήτε δεν στέρισαν τον πολίτη από την παραλία, ε, έχτισαν στο εσωτερικό της γης. Δεν ήταν ένας ευαίσθητος χώρος ζώνη, ήταν μια εσωτερική πεδιάδα, ιδιωτική ιδιοκτησία, με συγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο για την οικοδόμηση. Για την αναδρομικότητα του νόμου, η Πόρια Μπράβα εμφανίστηκε το 65 με το πρώτο χωροταξικό σχέδιο. Το σχέδιο πρόσβαση προς τη θάλασσα 1968. Ορισμός του θελάσσιου χώρου το 1970 στην παραλία. Με βάση αυτή τη γραμμή έχει γίνει η καταγραφή των οικοπαίδων και ο Λέιντε Κώστα, νόμος των ετών, ψηφίστηκε 20 χρόνια μετά. Η νέα τροποποίηση της οριοθετικής γραμμής του 2008, ακόμα 20 χρόνια μετά, δηλαδή 40 χρόνια μετά που άρχισαν να πολλούνται τα τεμάχια αυτά γης και την καταγραφή στο κτηματολόγιο. Το κράτος λέει ότι είναι συνταγματικό. Οι πρώτες κατασκευές έγιναν το 1965. Ο πρώτος νόμος ψηφίστηκε το 1978. Υπήρχε πάνω από 10 χρόνια πριν από τον Ισπανικό νόμο. Μια χώρα δεν μπορεί να αρνηθεί την ιστορία της, πρέπει να ενσωματώνει την ιστορία της και το παρελθόν της. Ας ξεχάσουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Βέβαια, η Ισπανία χρειάστηκε να προσαρμοστεί στη δημοκρατία, να μπει στην κοινή αγορά, να μπει στην Ευρώπη, να προσαρμοστεί στο ευρώ. Όλα τρέχανε και βιαζότανε. Μπορεί να γίνανε και λάθη λόγω αυτού, αλλά δεν πρέπει να αρνηθεί το παρελθόν. Δεν είναι σωστό να πληρώσει ο ιδιώτης, ο πολίτης, τα σφάλματα και την έλλειψη ελέγχου εκ μέρους των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το κράτος μας λέει υπεύθυνοι είναι οι συμβολογράφοι και οι υποθηκοφύλακες. Το κράτος όμως τώρα ζητάει την αλλαγή του κτηματολογίου και ορίζει τη νέα γραμμή για τον υγειαλό. Πώς είναι δυνατό να οριστεί μια γραμμή η οποία δεν είχε οριστεί από το κράτος στο παρελθόν. Και ήταν ευθύνη του κράτους να έχει οριστεί μια τέτοια γραμμή ευθύ εξ αρχής. Ορισμένες αρμοδιότητες δόθηκαν στην Καταλωνία. Πώς μπορεί ο πολίτης να αμφισβητήσει το κοινοβούλιο, τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου της Καταλωνίας, σοβαρέ οι οικονομικές επιπτώσεις. Έχει σταματήσει να λειτουργεί η τοπική οικονομία. Καθένας δεν θέλει να επενδύσει σε ένα αγαθό το οποίο κινδυνεύει νομικά. 40% ανεργία νέων. Είναι λογικό να βασβητηθεί η αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων, η εμπιστοσύνη στην αγορά. Οι ιδιοκτήτες μιλάνε στις εφημερίδες, απευθύνονται στα προξενία και τώρα που χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη για την οικονομική ανάπκαμψη θεωρούμε ότι πρέπει να μιγήσει και η Ευρώπη. Στην Εμπούρια Μπράβα δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Επί 40 χρόνια δεν είχαμε πλημμύρες λόγω καλού προγραμματισμού. Το... Υπάρχουν ατομικά σπίτια χτισμένα ατομικά, γιατί να δεχθούμε την απαλουτρίωση τη στιγμή που έχουν χτιστεί νόμιμα, ενώ ταυτόχρονα παραδίπλα χτίζονται νέα χωριά με τεράστια οικοδομήματα για χιλιάδες άτομα. Πλήττονται οι πολίτες που σεβάστηκαν, που τήρησαν τους κανόνες και ανεχόμαστε, ανέχονται μάλλον, την κυροδοσκοπία. Μας μιλάνε για το γενικό συμφέρον που πρέπει να υπερισχύσει του ατομικού συμφέροντος. Αλλά το γενικό συμφέρον για να εξασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη, δεν σημαίνει σεβασμός του ατόμου και σεβασμός της κατοικία του. Γι' αυτό το δικαίωμα διεκτησίας, εφόσον η αγορά είναι νόμη, δεν είναι ένα καπρίτσιο ενός ατόμου. Αν δεν υπάρχει εγγύηση τάξης, θα έχουμε ή αναρχία ή δικτατορία. Γι' αυτό το, ο σεβασμός του δικαίωμα της κατοικίας είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Γι' αυτό πρέπει να τύχει σεβασμού το κτηματολόγιο που είναι η μόνη εγγύηση αυτής της ιδιοκτησίας. Προτείνεται αποζημίωση με μορφή προσωρινής παραχώρησης. Δηλαδή, ξόδεψε κανείς, δούλεψε, εξοικονόμησε για να αγοράσει και τελικά είναι ενοικιαστής του σπιτιού του. Αν δουλεύεις έχει χρήματα να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Είναι λογικό να είσαι ενοικιαστή του αυτοκίνητου αυτού για 5, 10, 20, 50 χρόνια όσο αποφασίσει το κράτο. Φυσικά μπορεί να ζήσει κανεί με κατάσταση leasing. Το κάνουν μερικέ χώρε. Αλλά οι κανόνε του παιχνιδιού έπρεπε να είναι σαφεί από την αρχή και όχι να αλλάξουν καθοδόν. Διότι η εργασία και η προσπάθεια για την αγορά δεν είναι ίδια. Γι' αυτό ζητούμε να χρησιμοποιήσετε ό,τι επιρροή έχει τη Ισπανία να προτεθεί μια παρέμβαση, μια διαπραγμάτευση με διαιτησία μέσω ε, επιτρόπου της Ευρώπης. Την αφορά την Ευρώπη αυτό. Εμείς προσπαθούμε πάση θυσία, προκειμένου η κυρία Σπινόσα που είναι αρμόδια για αυτό, η κυρία Σάλγκαντρο που είναι η, η Υπουργό Οικονομία ή και ο κύριος Θεμπατέρα ο ίδιος να αναθεωρήσουν και να μελετήσουν κατά περίπτωση το νόμο αυτό περί Αιγιαλού, έτσι ώστε να υπάρχει σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή σεβασμός μέσω του κτηματολογίου, της ιδιοκτησίας και των συμβολογραφικών πράξεων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, παρακαλώ και πάλι τους αναφέροντες να είναι σύντομοι. Είμαστε ούτε καν στο 50% των αναφερόντων και μας μένει μία ώρα το πολύ. Μαργαρίτα Γκαρσία Χάιμε Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η περίπτωσή μας είναι η περίπτωση εννέα οικογενειών που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που εθίγησαν από έναν κακό νόμο, έναν άδικο νόμο που δεν σέβεται το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση εδώ για να πω στον κύριο Μαρτίνες ότι αν έχετε την ίδια αντίληψη περί ιδιωτικών δικαιωμάτων ή ατομικών δικαιωμάτων με αυτές που έχει το καθεστώς του κάστρο, τον κάστρο μάλλον, εντάξει, το καταλαβαίνω. Υπό αυτό το πρίσμα το δικαίωμα ιδιοκτησίας ιδιωτικής δεν ένοιξε θεμελιώδη δικαιώματα. Το 1980, πολύ πριν δηλαδή τον ε, νόμο του 88, κατασκευάσαμε νόμιμα με έγκυρες απολεδομικές άδειες και δομικές άδειες τα σπίτια μας. Είχαμε ακόμη και την άδεια από τη διοίκηση των ακτών και μάλιστα οι αγορές αυτές έγιναν με δικηγόρους και με συμβολιογραφικές πράξεις. Η... Ε, έγινε και μεταγραφή των ιδιοκτησιών μας ως νομίμων και ιδιωτικών. Το 1990 η οριοθέτηση που έγινε από τον νόμο των ακτών χαρακτήρισε με νέο τρόπο την διαγράμμιση και πέρασαν οι δικές μας κατοικίες στο, στη δημόσια περιουσία και μάλιστα με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, με δόλιο τρόπο όμως, χωρίς να ενημερωθούν προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι κατά παράβαση του δικαίου και μάλιστα τελείως τυχαία μάθαμε για την νέα οριοθέτηση και προλάβαμε την τελευταία μέρα να υποβάλουμε τις προσφυγές μας. Το 2004 και μετά από 14 χρόνια διοικητικού αγώνα, με έγγραφα, ισχυρισμούς, ε, ε, τεκμήρια, δικαστικές πραγματογνωμοσύνες κτλ. Το ανώτατο δικαστήριο έβγαλε απόφαση υπέρ της διοίκησης, κηρύσσοντας επίσημα το κράτος ιδιοκτήτη των δικών μας κατοικιών. Παρ' όλα αυτά δεν απαλλασσόμαστε από την καταβολή του φόρου του περιουσίας, ούτε από την αποπληρωμή της υποθήκης μας. Και μάλιστα εξεπλάγει γιατί το όνομά μου δεν υπήρχε πια στο κτηματολόγιο. Αναφέρεται στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτήτης του σπιτιού μου το κράτος. Ο νόμος περί Αγιαλού ε, προβλέπει ως μοναδική αποζημίωση μία διοικητική παραχώρηση 30 ετών που μπορεί να παραταθεί θεωρητικά για, άλλα μια, για άλλη μία 30 ετία. Δυστυχώς όμως ε, αυτό προηγείται ε, της ανάκτηση, η, η, ανάκτηση μάλλον της περιουσίας προηγείται της διοικητικής παραχώρησης. Δηλαδή το κράτος θα μας κάνει έξωση από τις κατοικίες μας χωρίς να προβεί σε αυτή την παραχώρηση. Και μάλιστα οι παραχωρησει αυτε αυτές έχουν αξία 10-20.000 ευρώ το πολύ. Επίση, έχουμε την κατασκευή μια πλακόστρωση λωρίδα παραλίας πολύ αμφίβολη χρησιμότητα που δεν τη ζήτησε ο κόσμο, απλώς δίνει δίνει έναν χαρακτήρα πεζοδρόμηση στην παραλία και θα την φορτώσει με τόνους τσιμέντου, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία χωρίς ε, καμία τέτοια ανάγκη πλακόστρωσης. Πώς ισχυρίζεται η Ισπανική κυβέρνηση ότι προστατεύει το περιβάλλον. Άλλωστε, μετά την δημοσίευση του νόμου έχουν εγκριθεί πάρα πολλά ε, οικονομικά σχέδια αστικής ανάπτυξης ε, αμφίβολης περιβαλλοντικής ε, συμβατότητας. Ενώ εμείς ενημερωθήκαμε για την πρόταση κατεδάφισης των ε, οικειών μας. Καταγγέλουμε την τον αυθαίρετο χαρακτήρα της οριοθέτησης, χωρίς προκαθορισμένα τεχνικά κριτήρια. Φύγει ορισμένου η νέα οριοθέτηση, ενώ σέβεται άλλους, παρόλο που βρίσκονται στην ίδια απόσταση από τον Αιγαλό Υπάρχει σαφή ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων συγκροτημάτων εις βάρος των απλών πολιτών. Προστατεύονται τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ενώ καταστρατηγούνται τα συμφέροντα των πολιτών. Ο νόμος αυτός έχει μοναδικό στόχο να δημεύσει τις περιουσίες από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Πρόκειται για ένα νόμο που στηρίζεται σε μια χαλαρή δικαιοσύνη η οποία αποφασίζει υπέρ της διοίκησης ε, στα 96,7% των περιπτώσεων δημιουργώντας μια, δημιουργώντας μια τεράστια αβεβαιότητα δικαίου. Πρόκειται για ένα διαστραμμένο νόμο και στα 22 χρόνια εφαρμογής του ο νόμος αυτός δεν εξυπηρέτησε τις υποτιθέμενες προθέσεις διαφύλαξης των ακτών και του υγιαλού. Γιατί ε, στην περίοδο αυτή είχαμε τη μεγαλύτερη αστική ανάπτυξη στις Ισπανικές ακτές. Είναι λοιπόν ένας αποτυχημένος νόμος και ένας νόμος που προβλέπει αναδρομική ισχύ και εφαρμογή του, καταστρατηγώντας νόμιμα δικαιώματα κυριότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί συνταγματικό. όσο και αν το δικαστήριο ισχυρίζεται ότι είναι συνταγματικό. Είναι αντισυνταγματικό αυτό ο νόμος, γιατί καταστρατηγεί και το κοινοτικό δίκαιο, αλλά παραβιάζει και το ίδιο το Ισπανικό Σύνταγμα. Θα ήθελα να παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να εμποδίσουν σε ένα κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει ένα τέτοιο διαστραμένο νόμο, όπω είναι ο νόμο περί που μάλιστα κατάφορα και χονδροειδώς παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει να υποχρεωθεί η Ισπανική κυβέρνηση να μεταρρυθμίσει αυτό το νόμο προκειμένου να σεβαστεί τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών όπως κατοχυρώνονται στον θεμελιώδη χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στοιχειωδών θεμελιωδών ελευθεριών. Επίσης θα πρέπει να τηρηθεί η συνθήκη της Λισαβόνας ό,τι αφορά τη μη αναδρομική εφαρμογή του νόμου και στην ανάγκη δίκαιη αποζημίωση σε περίπτωση απαλωτρίωση. Σας ευχαριστώ. Grazie Καλημέρα. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Χθε ήμουνα παρόν κατά τη δήλωση της Ισπανικής Αντιπροσωπείας για τον νόμο περί Αιγιαλού. Επίσης ήμουνα εδώ πέρσι το Ιανουάριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανική Αντιπροσωπεία που κατέστησε τόσο σαφές γιατί υπάρχουν τόσα προβλήματα με τον Ισπανικό νόμο περί Αιγιαλού Ποιε είναι οι ευαισθησίε που υπάρχουν εδώ πέρα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με ένα από τα βασικά οικονομικά σκάνδαλα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ε, στην αναφορά 119 που αφορούν την εφαρμογή του, του ε, Ισπανικού νόμου περί Αγιαλού. Προσπάθησα θα προσπαθήσω να σας ε, παρουσιάσω στα πέντε λεπτά που έχω ε, την ε, λειτουργία του Ισπανικού νόμου περί Αιγελού και που ουσιαστικά υπό άλλες συνθήκες θα θεωρεί το εγκληματική δραστηριότητα. Εγώ μένω στη Βέρα Πλάγια, η οποία καταστρέφεται από έργα της Ισπανικής Διοίκησης. Μπορεί να χάσω το σπίτι μου και το βιός μου. Ένα από τα έργα ε, το έργο που έχει να κάνει με την ανάκτηση των ακτών ανάμεσα στο, ε, στον ποταμό Αρμανζόρα και το ε, λιμάνι της Γκαρούτσα πρώτη φάση πραγματοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παρά τις αναφορές που έχουν γίνει, είχε, είχαν ακουστεί προειδοποιήσεις σχετικά με την διάβρωση των ακτών. Τίποτα όμως δεν έγινε. Ε, οι νέες συνθήκες ε, ε, ωφέλησαν ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται βόρεια από μας. Παρότι αρχικά το ξενοδοχείο αυτό βρισκόταν πολύ πιο κοντά αρχικά στην ακτή από ότι οι δικές μας ιδιοκτησίες. Δεν χρειάζεται να σας, να σας δώσουμε εξηγήσει σχετικά με τη διάβρωση αυτή. Η πρώτη φάση αυτού του εξαιρετικού έργου ε, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι όλη η περιοχή μας ε, θα ενέπιπτε στην, ε, στον Ισπανικό νόμο περί γυαλού και ότι η επίθεση κατά της ιδιοκτησίας μας θα λόγω της τεχνητής ε, διάβρωσης ε, θα ε, δικαιολογείται από τον νόμο. Ο νόμος αυτός επιτρέπει στο Ισπανικό κράτος να κατασχέσει οποιαδήποτε περιουσία τώρα, στο παρελθόν, στο μέλλον που, και λόγω φυσικών ή τεχνητών συνθήκων. Και ακριβώς εδώ είναι το πρόβλημα. Εγώ βλέπω να, να διαβρώνονται οι ακτές, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση από ε, το σχετικό Υπουργείο. Ε, στο φάκελο θα βρείτε ε, επιστολή μου προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, την κυρία Σπινόζα. Δεν έλαβα καμία απάντηση. Επίσης, στα δικαστήρια έχω προσφύγει επανειλημμένα, δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει λύση να αποτραπεί ο κίνδυνος ε, για τις κατοικίες μας ε, ή τους κοινού χώρους. Υπάρχει πολύ απλή απάντηση. Όλα περιέχονται στην αναφορά αυτή και οι υπεύθυνοι έχουν ε, τα θέματα αυτά στο γραφείο τους. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Η επέκταση του, της, της Μαρίνας της ε, Καρούτσα θα έπρεπε να ε, ε, ολοκληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο και θα έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της, του προγράμματος ανάκτησης των ακτών. αυτό έχει ζητηθεί πολλές φορές προτού η, ζημιά να, να μην μπορεί να διορθωθεί πια. Ε, η ε, αποκατάσταση των ακτών είναι κάτι εύκολο, φθηνό, ε, περιβαλλοντικά και τουριστικά η καλύτερη λύση και θα έπρεπε να γίνει. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ευθυγραμμίζεται με την πολιτική κατάσχεση της παρούσας κυβέρνησης. το ότι λένε ότι οι ακτές μπροστά τα σπίτια μας διαβρώνονται λόγω της φυσικού φαινομένου, αυτό είναι γελίο αυτό που βλέπουμε είναι η Ισπανική διοίκηση, η Ισπανική κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τον, λόγο τον νόμο αυτόν για να πετύχει τα αποτελέσματα που θέλει. Τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι νόμιμα, αλλά εμείς αμφισβητούμε την νομιμότητα του νόμου αυτού. Αμφισβητούμε την πρόθεση μιας ε, δημοκρα... Ε, αμφισβητούμε τις προθέσεις ε, της δημοκρατικής αυτής κοινωνίας Αμφισβητούμε το επιχείρημα περί κοινού συμφέροντος ε, της ε, ισπανικής κυβέρνησης. Τα συμφέροντα που διακυβεύονται είναι τεράστια. Πρέπει να αναγνωριστεί αυτό. Πολλά, πολλές κατοικίες θα επηρεαστούν, χιλιάδες σπίτια θα επηρεαστούν και ε, το κράτος θα έχει αποκλειστικότητα στην ιδιοκτησία του, των ακτών. Μιλάμε για πολλά χρήματα και όπως ε, στη παράδειγμα της Βέρα Πλάγια με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται μια στρατηγική που καλύπτεται από τον νόμο περί για να ε, αφαιρέσει από τους ε, ανθρώπους τα νόμιμα συμφέροντά τους. Ο νόμος περί είναι ένα μέσο, ένα όπλο θα λέγαμε, με αμφισβητούμενους στόχους. Ε, αποτελεί αντίφαση η Ισπανική κυβέρνηση να εφαρμόζει τον νόμο αυτόν ε, αναδρομικά και να μην προστατεύει τους δημόσιους χώρους και τους πολίτες όπως είναι η υποχρέωσή της σύμφωνα με τους δημοκρατικούς κανόνες ε, της συνταγματικής φιλοσοφίας. Επίσης, η ανταλλαγή ιδιοκτησίας με περιορισμένη παραχώρηση είναι κάτι απαράδεκτο θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη και σωστή αποζημίωση. Ε, αυτό απαιτείται από τη δημοκρατία. Αλλά με τον νόμο αυτόν ε, αυτό δεν γίνεται. Το κράτος επένδυσε στις ε, τζάμπα και μιλάμε για νομική αβεβαιότητα, διάκριση, ε, αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι υπερβολικά πολλά αυτά για πέντε λεπτά. Αυτό που συμβαίνει στη Βέρα Πλάγια ε, είναι παράδειγμα όλων αυτών. Και εφόσον χρησιμοποιήθηκαν ε, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελπίζω αξιότιμα μέλη της Επιτροπής να θεωρείτε και γι' αυτό ζητώ να δείτε θετικά την ε, αναφορά 119 και όλες τις αναφορές ε, που έχουν παρουσιαστεί από τους ε, ανθρώπους που απειλούνται από τις Ισπανικές αρχές λόγω του νόμου του Αγιαλού. Θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί Αγιαλού και οι σχετικές διατάξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Αντώνιο Λουίς Γκαρσία. José Antonio Luis García. Είστε ο κύριος Χωσέ Αντώνιο Λουίς Γκαρσία. Είμαι ο εκπρόσωπος του Χωσέ Αντώνιο Λουίς Γκαρσία εκεί είμαι ο Τομάς Γκονσάλες Δία, αναφέρον ε, για την περίπτωση του Τσόβιτο. Πώς είπατε ότι λέγεστε Τομάς Γκονσάλες Δία. Είμαι αναφέρον για το Τσοβίτο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία, τη μοναδική ευκαιρία που έχουμε κάθε πέντε χρόνια μας ζητάτε την ψήφο μας. Για πρώτη φορά ζητούμε και εμείς κάτι από εσά να μας ακούσετε στην Επιτροπή σας είδατε ότι έχετε στην ημερήσια διάταξη πληθώρα αναφορών από πολλά σωματεία και ενώσεις και ομάδες με εκπλήση που δεν υπάρχει ούτε ένας ξενοδόχος που να ζητά προστασία της Επιτροπής Αναφορών για να μην καταδεφιστεί το ξενοδοχείο του που βρίσκεται στις Ισπανικές ακτές. Έχουμε αλλάξει άρθιν την ε, ομιλία μας, προσαρμόζοντάς τη ε, στις χθεσινές δηλώσεις ε, της κυρίας Αλήσια Δεπάς, που στις 8 Οκτωβρίου προκάλεσε πόλεμο στο Τσοβίτο που είναι μια, ένας ψαράδικος οικισμός ε, στα Κανάρια νησιά. Εκεί καταπατήθηκαν όλα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και μάλιστα ε, μας αποκαλούν παράνομους και το ψαροχώρι του Τσοβίτο πληρώνει φόρους. Εκεί όταν πληρώνουμε φόρους είμαστε νόμιμοι. Είμαστε παράνομοι μόνο όταν ε, αποφασίζουν να καταδαφίσουν τα σπίτια μας. Πολλά αναφέρθηκαν για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι δικαίωμα, τι ανθρώπινο δικαίωμα τηρήθηκε από την Ισπανική κυβέρνηση. Αν δείτε εικόνες ε, πώς ε, αντιμετωπίστηκαν οι πολίτες του Τσοβίτο, που το μοναδικό έγκλημα που διέπραξαν είναι να είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διαπιστώσετε πως εξευτελιστικά μας μεταχειρίστηκε η Ισπανική κυβέρνηση. Μια υποτιθέμενα δημοκρατική κυβέρνηση που μάλιστα χθες με πολιτικούς εκπροσώπους της αρνήθηκε την συμπερίληψη της ατομικής ιδιοκτησίας στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε απλώς πολίτες. Εδώ καταστρατηγούνται όλα τα, τα άρθρα του Ισπανικού Συντάγματο. Καταστρατηγείται η Συμφωνία του Άρχου, η Συνθήκη τη Λισαβόνα. Χρειάστηκε να έρθουμε μέχρι τι Βρυξέλλε. Είδαμε και ακούσαμε χθε ε, σχεδόν σε όλε τι ε, παρεμβάσει ε, με εξαίρεση μία, ότι είναι δίκαιος ο νόμος που περιέγει αλλού. Ο νόμος που εφαρμόζεται μόνο στους πιο αδύναμους, που δεν βλέπει ένα τεράστιο ξενοδοσιακό συγκρότημα που αναγείρεται στη Βίγια Πεσόα στη Γαλλικία. Εθελοτυφλοί όταν κτίζονται τεράστια ξενοδοχεία και καταστρέφονται εικόνες των ακτών. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε εδώ ξενοδόχους, γιατί για τους ξενοδόχους υπάρχουν κενά και παραθυράκια στον νόμο. Εδώ πολλά αναφέρθηκαν ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε να υποβάλουμε τις προσφυγές μας για την οριοθέτηση της ακτής της Τενερίφης μέχρι το Υπουργείο. Και συγχαίρω την Αλήσια Δεπάς που χθε ε, ήρθε να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες. Αλλά αντιμετωπίζω τις κατηγορίες δεν σημαίνει να έρθω απλώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 8 με 10 χρόνια ζητούμε από το Υπουργείο ακρόαση και δεν έχουμε γίνει δεκτοί το τσοβίτο δεν ε, καταστρέφεται ή δεν καταταφίστηκε γιατί παραβιάζει το, το νόμο περί Αγιαλού, αλλά γιατί αυτό που ενδιαφέρει την Ισπανική κυβέρνηση είναι μόνο αυτό που βρίσκεται μπροστά στο τσοβίτο, που είναι μια μαρίνα αναψυχής. Και το πίσω τμήμα του τσοβίτο ε, που απαρτίζεται από ψαράδικους οικισμούς παραδοσιακούς και που είχε πράσινη, πράσινη ζώνη και πάρκο ε, ενδιέφερε μόνο για το οικόπεδο για να δημιουργήσει πολυτελής επαύλης. Οπότε δεν θέλει η Ισπανική κυβέρνηση φτωχούς δίπλα στους πλούσιους. Δίπλα στο Τσοβίτο έχουμε 16 με ή 18 πολυόροφα κτίσματα και οικόπεδα που έφαγαν ε, τον Αιγιαλό και τις ακτές της Τενερίφης. Αν δούμε τη νότια πλευρά της Τενερίφης, πιστώνουμε ότι έχουμε ξενοδοχειακά συγκροτήματα που βρέχονται από το νερό, με ιδιωτικές παραλίες. Με ιδιωτικές παραλίες. Εκεί είναι που καταπατάτε το δικαίωμα του πολίτη να πάει και να κάνει ελεύθερα μπάνιο οπουδήποτε στην Τενερίφη. Και αν δούμε την υπόλοιπη ακτογραμμή της Τενερίφης, πιστώνουμε ότι τρία τέταρτα των ακτών στο Λασαρότε, στην Φουέρτε Βεντούρα, στην Γκραν Κανάρια, και στην Πάλμα ίδια κατάσταση αντιμετωπίζουμε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, εμείς δεν είμαστε κατά του νόμου περί ακτών και γυαλού. Όχι. Είμαστε κατά της εφαρμογής του νόμου αυτού και της επιλεκτικής εφαρμογής του νόμου, γιατί αναφέρθηκε ως καινοτόμο ο νόμος. Για ποιο νόμος είναι καινοτόμο, εξαρτάται. Για ποιον εφαρμόζεται. Για μας πάντως σίγουρα δεν ήταν καινοτόμο αυτός ο νόμος. Εμείς ε, είπαμε ότι αν βλέπατε τις εικόνες ε, του Τσοβίτο, το πώς καταδαβίστηκε, ίσως αφυπνιζόταν κάποιες συνειδήσεις. Ήρθαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταδικάσετε κι εσείς την αυθαιρεσία και τη δίμευση ατομικής ιδιοκτησίας του βιού και του, της περιουσίας των πολιτών. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί αυτή η κατάσταση, να μην υπάρξει νέο τσοβίτο και πάνω από 400.000 άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από το νόμο αυτό ε, για τις ισπανικές ακτές. 23 από τα 31 σπίτια του Τσοβίτο έχουν καταδαφιστεί. Ελπίζουμε όμως να μην υπάρξει δεύτερο Τσοβίτο. Το ανθρώπινο δικαίωμα, όπως είπε χθε ε, ο κύριος Μαρτίνες, ε, δεν καλύπτει και το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας. Μήπως δεν διαβάσατε το άρθρο 17, κύριε Μαρτίνες, γιατί κάτι τέτοια λέει ο Τσάβες. Προτιμώ όμως το δημοκρατικό καθεστώς, όπως κατοχυρώνεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Grazie. Jimenez Domingo. Jimenez Domingo. Κυρία Ματζόνη. Ένα διαδικαστικό λέει ο κύριος Μπασινάρο. Παρακαλώ όλους τους αναφέροντες να μην κάνουν παρατηρήσεις για πολιτικούς σε σχέση με πολιτικού σχηματισμού ή πολιστικό χρώμα στην Επιτροπή μα. Πρόεδρος, σωστό. Παρακαλώ οι αναφέροντες να το τηρούν αυτό. Χιμένες Ντομίνγκο. Buenos días. Καλημέρα σα. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, ακολουθώντα τι συστάσει τη Προέδρου, θα κάνω θα προσθέσω και εγώ κάποιες πινελιές και θα κάνω μερικές τροποποίησεις στην αρχική μου ομιλία. Γιατί τη χθεσινή μέρα τη βίωσα ως επίθεση εναντίον μας. Δηλαδή, εμείς είχαμε αρχίσει να βαδίζουμε σε ένα δρόμο που αρχίζει και αποσαφηνίζεται από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Λόιτ θα λάβει από τους ψηφοφόρους του διάφορες πληροφορίες για να ενημερωθεί για την προθεσμία, γιατί θα ήθελα μετά το τέλος συνεδρίασης να μου πει αν έχει αλλάξει γνώμη ε, σε σχέση με χθε. Γιατί αν δεν έχει αλλάξει γνώμη θα έχουμε αποτύχει. Αν όμως έχει μετακινηθεί κάπως η γνώμη του σημαίνει ότι έχουμε προχωρήσει. Αφήστε τον πόντιο πύλα. Θα πρέπει να πάψουμε να ανήπτουμε τα σχήρας μας και να κάνουμε κάτι επιτέλους. Εγώ ανέφερα τον θεοδοσιανό κανόνα στην παρέμβασή μου που είναι ως λίθος ενός κράτους δικαίου. Εκεί αναφέρεται ότι δεν προβλέπεται αναδρομική ισχύ των νόμων. Όλα τα συντάγματα που σέβονται το όνομά τους περιλαμβάνουν μία παράγραφο που μεταφέρει ουσιαστικά αυτόν τον θεοδοσιανό κανόνα του ρωμαϊκού δικαίου, γιατί οι Ρωμαίοι επινόησαν το δίκαιο. Με βάση λοιπόν αυτό τον κανόνα της μη αναδρομικότητας, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τι συνέβη χθες εδώ, στην συνεδρίασή σας. Και συνεχίζοντας τις επιθέσεις, η κυρία Αλήσια Πας Αντολίν ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, γιατί μίλησε για ένα μεταβατικό, για ένα νομικό μεταβατικό καθεστώς. Δηλαδή, αυτό αντικαθιστά την αναδρομικότητα των νόμων τι μεταβατικό νομικό καθεστώς ισχύει στην περίπτωση αυτή. Ε, μεταβατική είναι η ζωή μας, γιατί έχει ένα τέλος. Και η δική μας και η της κυρίας Αλήσια Πάς. Αλλά αυτό το καθεστώς δεν είναι μεταβατικό. Γιατί ε, και η εκπρόσωπος ε, των ακτών, αυτή που φέρεται εκπρόσωπος των ακτών στον τύπο, σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό του Αλικάντε, είπε ότι είναι αρμόδιοι για πολλά χιλιόμετρα των ακτών. Διαβάστε την πρώτη παράγραφο της αιτιολογικής έκθεσης του, του νόμου περί που λέει ότι 7.850 χιλιόμετρα είναι το εύρος των ακτών, δηλαδή διπλάσιο από αυτό που ισχυρίστηκε η κυρία ότι αρμόδια, γιατί είπε 3.500 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Και αν περάσουμε στις μεταβατικές διατάξεις, γιατί εκεί είναι το ψαχνό της υπόθεσης, και από εκεί είναι που θα πρέπει να βρούμε το ζουμί, γιατί ο νόμος είναι σαν την πάντα του Δήμου. Ο νόμος είναι η μπάντα και η απήχηση, η ηχός που ακολουθεί την, την ορχήστρα είναι ο κανονισμός. Ένας πρόδρομος του κ. Μαρτίνες και μάλιστα δεν ξέρω γιατί δεν κάθεται στο Προεδρείο, ο κύριος Ρομέρο Ροβλέδο, πρόδρομος του κύριου Μαρτίνες, ψηφοθύρας γνωστός ε, που πλήρωνε 3-4 ε, τρει-τέσσερι πεσέτες για να αγοράσει ψήφου. είπε, ε, είχε πει τότε την περίφημη φράση «Κάντε εσείς τους νόμους και αφήστε σε μένα τους κανονισμούς». Τι να κάνουμε με τον νόμο που έχει δέκα άρθρα, που κρίθηκε μάλιστα συνταγματικό από το συνταγματικό δικαστήριο. Αν στη μέση ενός άρθρου διαγράφεται μία παράγραφος και ερμηνεύεται, η... έχουμε κανονισμό που τον εφαρμόζει όπως έτσι, έχουμε... αν έχουμε ένα φαγητό κατσαρόλας, ε, τι θα γίνει αν δεν βάλουμε αλάτι. Τίποτα. Θα είναι άνοστο, αλλά μπορεί να είναι και υγιεινό. Ε, μπορούμε όμως από το βραστό να βγάλουμε και το κοτόπουλο. Γιατί πρέπει να σκοτώσουμε και την κότα. Ε, ας βγάλουμε και το χοιρινό, γιατί έχει χολυστερίνη. Ας μην βάλουμε και τα ρεβίθια στο βραστό μας. ας μην βάλουμε και το νερό. Ε, τι βραστό, τι φαγητό κατσαρόλα είναι αυτό αφού έχουμε αφαιρέσει όλα τα συστατικά. Τι νόμος είναι αυτό αφού το, το δικαστήριο έχει αφαιρέσει ένα σωρό άρθρα και παραγράφους. Είναι συνεκτικός αυτός ο νόμος, εξακολουθεί να θεωρείται νόμος. Ή όταν ε, εφαρμόζεται ένας εκτελεστικός ε, κανονισμός 200 και άρθρων, πώς θα το παρακολουθήσουμε, πώς θα εντοπίσουμε τις αντιφάσεις του. Εκεί που λέει άσπρο εννοεί μαύρο, και όταν σταματήσουν όλα αυτά, τι έχουμε, μας μένει μια λευκή σελίδα ή μας μένουν ελάχιστες διατάξεις. Εντάξει, είναι ιδιότροπη η φύση, αλλά η ανθρώπινη φύση είναι ακόμη πιο ιδιότροπη. Και αν είναι κανείς τόσο ε, λεπτολόγος κομμουνιστός, ε, κομμουνιστής από τον κύριο Μαρτίνες, ε, είναι το αποκορύφωμα. Βλέπετε την ακτογραμμή. Η ακτογραμμή μπορεί να τροποποιείται. Μπορεί να, να τροποποιείται και η προστατευόμενη απόσταση από την θάλασσα έχουμε απόσταση από 5 μέτρα ενός πεζόδρομου για παράδειγμα, ενός ε, μονοπατιού, από 5 μέτρα ενός ε, μονοπατιού μπορεί να είναι η απόσταση αν πρόκειται για ξενοδοχείο. Διαδικαστικό. Από τον κύριο Μάγερ, διαδικαστικό. Θα να παρακαλούσα τους ετούντες να περιοριστούν στο δικό τους ζήτημα, στη δική τους αναφορά. Γιατί αν θέλετε όντως να μιλήσετε για το θέμα σας, πολύ ευχαρίστως. Αν όμως συνεχίσετε τους προσωπικούς επενιγμούς κατά συγκεκριμένου βουλευτή, τότε παρεκτρεπόμαστε από τη συζήτηση. Σας θέρμο παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε στην αναφορά, αν όντως αυτό σας ενδιαφέρει. Μα το θέμα μας λέει είναι ο, ο κύριος τότε αποφύγετε τους υπενιγμού και τα υπονοούμενα για συγκεκριμένο ευρωβουλευτή. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Έλμερ που χθε ένα συμπολίτη μου το κατηγόρησε και του ζητώ συγγνώμη. Πιστεύω ότι υπάρχει ελευθερία έκφραση εδώ. Αν τώρα μου στερείτε το λόγο, τι να πω, τι ελευθερία έκφραση είναι αυτή. Λοιπόν, μέσα στου κανόνε, τι προβλέπει ο κανόνα, ότι αν είναι υπερπολιτελέ το ξενοδοχείο, η προστατευόμενη απόσταση είναι 5 μέτρα από, την από, την, από το νερό, από τη θάλασσα. Αν είναι ένα απλό πολίτη, μπορεί να είναι 20 μέτρα η προστατευόμενη ζώνη. Αν ενδιαφέρει μια περιοχή, μπορεί να είναι 100-200 μέτρα, γιατί μπορούμε να αφαιρέσουμε την περιουσία και ενό εχθρού μα. Γιατί να μην γίνει και και 200 μέτρα η προστατευόμενη ζώνη. Αυτά είναι τα καπρίσια της οριοθέτησης που εφαρμόζεται πολύ αφήσιμα και αυθαίρετα. Τι θα πει δημόσιο κτήμα ε, θαλάσσιο και χερσαίο ή αιγιαλός ή ακτογραμμή. Μέχρι που φτάνει. Φτάνει μέχρι το κτηματολόγιο μερικές φορές αυτή η προστατευόμενη ζώνη. Μπαίνει κανείς με, με την πουλντόζα και ζητάει και τα έξοδα της κατεδάφισης. Όλοι έχουμε κινητό. Ας κάνουμε μία μικρή άσκηση. Όλοι ακτιμούμε το κινητό μας για πολλές και διάφορες ιδιότητες. Τώρα βγαίνει, εκδίδεται ένας νόμος που λέει όχι, τα κινητά είναι κρατικά. Και από τη στιγμή που θα, τα κινητά θα γίνουν κρατικά, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του κινητού. Παρ' όλα αυτά τον πληρώνουμε εμείς. Απαλωτριώνει λοιπόν τα κινητά το κράτος και μας αφήνει τη χρήση του κινητού μόνο για το επόμενο δίμηνο. Στο μέλλον όμως, εμείς θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς ε, προς, τη... προς τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας, αλλά μετά από δύο μήνες το κράτος θα μας αποσύρει τα κινητά. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μία φράση του Θερβάντες που είπε ότι η ελευθερία είναι από τα πολυτιμότερα αγαθά που πήραν οι άνθρωποι από τους θεούς. Και στην Ισπανία, ελάτε να το δείτε με τα μάτια σας και να το εξηγήσετε, αυτή η ελευθερία διακυβεύεται. Ευχαριστώ. Ruth Martin Λένερτ, Τρία λεπτά. Μετά από τρία λεπτά θα σας διακόπτω. Γιατί πάνω από μία ώρα συζητάμε και δεν θα έχουμε χρόνο να τους ακούσουμε όλους. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ στην Επιτροπή σας και που έχουμε τη δυνατότητα να αναφέρουμε το πρόβλημά μας. Ε, και εμείς από την Αμπούρια Μπράβα ε, είμαστε. Ε, θα είμαι σύντομη όμως καθότι η κυρία Χόφμαν παρουσίασε ε, ενδελεχώς το θέμα. Η απαλωτρίωση γίνεται με τρομερό τρόπο, χωρίς καμία προσωπική κοινοποίηση και το 60% της περιουσίας μας επηρεάζεται. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε την, την ε, περιουσία μας. Ε, αυτό σημαίνει ότι χάσαμε την περιουσία μας στη Γερμανία επειδή ε, την πουλήσαμε για να αγοράσουμε το ακίνητό μας στην Ισπανία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα επιχειρήματα. Τα κανάλια ήταν πάντα κοινοκτήμα, ήταν πάντα δημόσια, ήταν πάντα ανοιχτά στο κοινό. Ε, η εισαγωγή στο κτηματολόγιο ήταν για μας η μεγαλύτερη δυνατή νομική βεβαιότητα και υπάρχουν, υπάρχει εδώ και 30 χρόνια ε, η περιοχή αυτή και θα έπρεπε να μπορούμε να, ε, να πιστέψουμε σε αυτό. Για μας τίθεται το θέμα τι, τι σύμβαση μπορεί να υπογράψει πια κανείς, τι είναι νομική βεβαιότητα. Διότι όλα είναι δυνατά τώρα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον ε, νόμο, το, η ζώνη των 6 μέτρων μπορεί να επεκταθεί στα 20 μέτρα. Γι' αυτό, κυρίε και κύριοι, έχουμε ε, απευθυνθεί σε εσά, διότι έχουμε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε να μα βοηθήσετε στην υπόθεσή μα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Grazie Kohler. C'è? Ah ja, okay. Liebe Abgeordnete, danke, dass ich... Αξιότιμοι βουλευτές, ευχαριστώ που μπορώ να πάρω το λόγο σήμερα. Θέλω να μιλήσω για τις ανησυχίες μας λόγω ενό μικρού σπιτιού που έχουμε στο μικρό ε, νησί των Βαλιαρίδων, Φορμεντέρα από το 1990 ε, έχουμε συνέχεια προβλήματα. Η Εσκριτούα μας ε, από το 1984 έγινε σύμφωνα με όλους τους κανόνες που αφορούν το κτηματολόγιο. Και στην Φορμεντέρα δεν υπάρχει υπερβολική οικοδόμηση ένα κτίριο επιτρέπεται να φτάσει το πολύ ε, στο ύψο ενό δέντρου. Δεν έχουμε οικοδόμηση στι ακτές ε, με εξαίρεση τα μεγάλα ξενοδοχεία για τα οποία, στα οποία θα αναφερθώ αργότερα. Ε, κάθε μέτρο ακτής μπορεί να είναι προσβάσιμο από όλους. Μπορεί κανείς να κάνει το γύρο του νησιού με τα πόδια. Στην Φορμεντέρα έχουμε ε, σεβαστεί πάντα τους ε, κανόνες της προστασίας των ακτών. Πολλοί ε, από εσά θα θεωρούν ότι η ζώνη των ακτών στην Ισπανία είναι 20 με 100 μέτρα. Εμείς απέχουμε 180 μέτρα από την ακτή και πίσω μας η οριοθέτηση Φτάνει τα 230 μέτρα. Ένα χιλιόμετρο πιο ε, ανατολικά η οριοθέτηση ε, φτάνει 350 μέτρα στα ιστορικά του νησιού και κάπου... Και αυτό σε σημείο όπου το νησί είναι, έχει ε, ε, πλάτος μόλις 1.400 μέτρα. Η Φορμεντέρα έχει 79 τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, έκταση ε, και το 13,2% περισσότερο από 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, έχουν απαλυτρωθεί από το, ανήκουν στο κράτος και αν προσθέσουμε και την δεύτερη ζώνη, την ζώνη των δουλειών, τότε χάνουμε το 30% των, της έκτασης του νησιού. 5 ε, με 6 χιλιόμετρα από το 1969 ε, έχουν ε, διατηρηθεί ως παρακτία ζώνη. πολλοί Ισπανοί και άλλοι αποκλείονται από τις ιδιοκτησίες τους. αγαπητοί Ισπανοί ευρωβουλευτές, ναι, θα ήθελα οι Ισπανικές οικογένειες να μπορούν να διατηρήσουν την κληρονομιά τους, αλλά και μεγάλοι κερδοσκόποι θα υποφεληθούν από την επέκταση τη ε, παρακτία ζώνης ε, από τα 5 στα 6 ε, χιλιόμετρα. Μου λένε ότι πρώην γερουσιαστής βρίσκεται μεταξύ των ιδιοκτητών των ξενοδοχείων και έχουμε τι μεγάλε αλυσίδε ξενοδοχείων Ρίου και Ινζοτέλ. Ερώτηση. τα μεγάλα ξενοδοχεία προστατεύουν καλά τις ακτές. Ε, επίσης, στον τίτλο 1, κεφάλαιο 1, άρθρο 4 του νόμου περί ακτών ε, αναφέρεται η κρατική παράκτια ζώνη ε, ως η ζώνη η οποία ε, φτάνει από την θάλασσα μέχρι, στο, μέχρι την κορυφή της παρακτής γραμμής. Αυτό των βράχων. Υπάρχουν όμως ε, βράχοι που δεν έχουν ε, ληφθεί καθόλου υπόψη. Υπάρχουν ε, βράχοι με ύψος 20 μέτρων που δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την οριοθέτηση. Κατά την οριοθέτηση στη Φορμεντέρα εν μέρη δεν έχει εφαρμοστεί το περιεχόμενο του νόμου. Κυρίες και κύριοι, το 1984 αγοράσαμε το μικρό μας σπίτι ε, εμπιστευόμενοι την ε, μελλοντική προσχώρηση της Ισπανίας στην ε, ευρωπαϊκή κοινότητα. Ελπίζαμε σε πρότυπα ιδιοκτησίας όπως αυτά που εφαρμόζονται στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη και κανένας από τους 40 ε, μικρούς ιδιοκτήτες ε, που, είναι γερμανικής, αγγλικής, ε, ολλανδικής, ιταλικής, ε, αυστριακής και ισπανικής εθνικότητας. κανένας από μας το 1988 δεν φαντάστηκε ότι σε, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαλωτριόταν η περιουσία μας χωρίς αποζημίωση. Ε, δεν μπορούσαμε ούτε να ε, ε, κληρονομήσουν τα παιδιά μας τις περιουσίες αυτές. Σε μια παραχώρηση μας δόθηκε μόνο. Με προπαγάνδα από στόμα σε στόμα ακούσαμε το 1990 σχετικά με την αναδρομική ισχύ του νόμου. Δεν λάβαμε ποτέ γραπτή κοινοποίηση, αλλά βρήκαμε την απαλωτρίωσή μας σε, σε, σε μια στίβα χαρτιά ε, στο Δημαρχείο ψάχνα, ψάξαμε μεταξύ πολλών ονομάτων στο όνομα Κούλερ και αυτή ήταν υποτίθεται η επίσημη κοινοποίηση και το πρόβλημά μας ε, είναι σχετικά μικρό όταν σκέφτομαι ε, τους άλλους ε, που επηρεάζονται. χτίζουν τις, τα, καταστήματα τους, τα καταστήματά τους, τα μικρά τους ξενοδοχεία. μιλάμε για δουλειά δύο-τριών γενεών η συνάδελφος Ρόζα ε, ε, Σταράς είπε ε, στις 8 Μαρτίου φέτος στο Στρασβούργο ότι ε, με, το, τις, ε, με το νόμο περιακτών το 70% των ε, τουριστικών εγκαταστάσεων θα εξαφανιστεί. Στην Φορμεντέρα όμως πάντα σεβαστήκαμε τους κανόνες για το περιβάλλον. Η κυρία Εσπινόσα, η Υπουργό Περιβάλλοντος της Ισπανίας, είπε τον Μάιο του 2008 ότι θα λυθεί το θέμα της Φορμεντέρα ως εξή, ότι θα επιτραπεί σε αυτούς που έχουν υποστεί απαλωτρίωση να χτίσουν ε, εντός ε, του ε, νησιού, με δικό τους κόστος βέβαια. Δεν υπάρχει όμως χώρος στο μικρό αυτό νησί να γίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα περιμένουμε η κυρία Εσπινόζα να βρει μια λύση κατά περίπτωση. Μιλάω και στο όνομα των κατοίκων του νησιού, θα το νιώθετε αυτό. Παρακαλώ, κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, κάντε κάτι ώστε ε, να έχουμε ε, μία νέα και δίκαιη οριοθέτηση, όπως μας την υποσχέθηκε ο κύριος Απατέρο τον Ιούλιο του 2009 κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Και παρακαλώ. επιτρέψτε φροντίστε να λάβουμε μια δίκαιη οριοθέτηση. Πότε θα τη λάβουμε αυτήν, πότε, πείτε μου. Αστρό. Τελευταία παρέμβαση, Δεκάστρο. Καλημέρα σας ε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Ονομάζομαι Χόνη του Ριβαρία και είμαι ο ιδιοκτήτης του Πόρτου Ερώτα, του Μήλου που βρίσκεται σε διαδικασία δίμευσης και ουσιαστικά ερήμωσης και καταστροφής από το τμήμα ακτών του Υπουργείου. Θα σας εξηγήσω τι συνέβη με το μήλο. Καταρχήν, το πιο προβληματικό σημείο του νόμου είναι η αναδρομικότητά του. Έχουμε εδώ σε αυτά τα έγγραφα που έχω στο χέρι μου και αυτά που βλέπετε στην οθόνη είναι επίσημα έγγραφα από το 1683. Και έχω εδώ στο τραπέζι όλα τα έγγραφα με τα βιβάσεις που έγιναν τους τελευταίους πέντε αιώνες και παρόλα αυτά δεν αναγνωρίζονται από το τμήμα ακτών. Χθες ε, η εκπρόσωπος της Ισπανικής Κυβέρνησης, η ε, Γενική Διευθύντρια των Ακτών, δεν ε, διευκρίνησε το ότι ε, η Ισπανία αναγνωρίζει ιδιωτικούς θύλακες ε, στη δημόσια περιουσία με βάση προηγούμενες νομοθεσίες όπως το νόμο περί υδάτων. Ο νόμος 8 παραβιάζει και την Ισπανική νομοθεσία που αναγνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων ιδιωτικών θυλάκων ακόμη και εντός της δημόσιας περιουσίας αρκεί να αποδειχθεί η ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας ή τίτλων κυριότητας όπως αυτοί, αυτούς που έχω εδώ μαζί μου. Ως εκ τούτου, ισχύει αναδρομικά από ό,τι φαίνεται ο νόμος περί αγιαλού. Ε, εμείς ισχυριζόμαστε ε, για την αναδρομικότητα, ε, ισχυριζόμαστε ότι ισχύει η αναδρομικότητα αυτού του νόμου, ότι εφαρμόζεται. Είναι σπάνιες ε, περιπτώσεις παλαιροϊκών μήλων στην Ισπανία. Τρεις έχουμε και μάλιστα και οι τρεις μήλοι χτίστηκαν με τον ίδιο τρόπο για να χρησιμοποιούν τα κύματα της παλήριας είναι κοντά στη θάλασσα. Και μάλιστα οι δύο ε, έχουν ε, εγκριθεί, αναγνωρίζοντα ιδιωτική περιουσία. Ο δικός μου όμω μήλος έχει δημευθεί, γιατί θεωρείται ότι περιλαμβάνεται σε δημόσιο κτήμα. Με τι σκεπτικό συμπεριλήφθηκε η περιουσία μου στην ε, κρατική περιουσία. Η μορφολογική μελέτη αναγόταν στον 17ο αιώνα. Ο δικός μου μήλος είναι από προηγούμενη εποχή. Θα έπρεπε η μελέτη που έγινε να κηρυθεί άκυρη. Άλλωστε, η ζώνη που αναφέρει ο, ο νόμος είναι 3 μέτρα, ενώ ο δικός μου είναι στα 2,48 μέτρα. Μάλιστα υπάρχουν τοπογραφικές μελέτες που αποδεικνύουν την ε, απόσταση του μήλου μου από την παραλία για πάνω από τρία μέτρα. Και μάλιστα η πραγματογνωμοσύνη που διέταξε το ίδιο το δικαστήριο αποδείχθηκε ότι έχω δίκιο εγώ. Ποια ήταν όμως η συνέπεια παρά την θετική γνωμοδότηση της πραγματογνωμοσύνης του δικαστηρίου και παρά το ότι η μορφολογική μελέτη ήταν μεταγενέστερη από τη δική μου αγορά, παρόλα αυτά ο μήλος μου χαρακτηρίστηκε κρατική περιουσία. Έχουν απαλωτριωθεί πολλά αγαθά. Για παράδειγμα, ο μήλο κατοικία, πάνω από 8.000 τετραγωνικά μέτρα αρρώσιμων καλλιεργειών, ε, με οποροκυπευτικά και σιτηρά. Και μάλιστα για πέντε αιώνε καλλιεργούν αυτά τα κτήματα. Και μάλιστα δημεύθηκε και το, το πιεστήριο του Μήλου που είναι 1,8 χιλιόμετρα πάνω από 18.000 τετραγωνικά μέτρα και το κτίσμα του Μήλου που θεωρήθηκε μνημείο από τον νόμο περί πολιτιστικής περιουσίας. Ο Μήλος Αθένιας που χαρακτηρίστηκε ιδιωτική περιουσία και η διαδικασία αγοράς και ανακαίνιση για να, να γίνει σαν το δικό μου αναγνωρίστηκε η αξία 3 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ εγώ τι λαμβάνω σε αποζημίωση από, τις ακτέ, από, τη... από τον νόμο περιακτών, τίποτα. Ο νόμος περιακτών και η Ισπανική κυβέρνηση δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση για την κατεδάφιση, την απώλεια της ιδιωτικής μου περιουσίας. Και κάτι που δεν είναι πειράζει εμένα, αλλά ολόκληρη την κοινωνία και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε για ένα ιστορικό μνημείο που έχει αναγνωριστεί ως πολιτιστική κληρονομιά. Πριν από ένα χρόνο είχαμε ένα, μια καταιγίδα στη χώρα των Βάσκων και μάλιστα σε ένα επίσημο έγγραφο της, του Τμήματος της ε, ε, ε, εκδόθηκε διάταγμα που με υποχρεώνει στην άμεση ανακαίνιση και επιδιόρθωση του μνημείου του Μήλου, ενώ ε, υπάρχει ένα αντιφατικό διάταγμα του τμήματος ακτών που με εμποδίζει να κάνω οποιοδήποτε διαδικασία επισκευή στο Μήλο. Βλέπετε ότι γίνεται ένας εκβιασμός γιατί το τμήμα ακτών δεν αναγνωρίζει την ιδιοκτησία μου και μου λέει ή θα δεχτείς να χάσεις την κυριότητά σου και να δεχτείς την παραχώρηση ή αλλιώς θα, θα γκρεμιστεί και θα, θα, ο μήλος. Υπάρχει άρθρο του, του Ισπανικού Συντάγματος που κρίνει αξιόπινη την δράση της, του τμήματος ακτών που ουσιαστικά οδηγεί σε φθορά ένα ιστορικό μνημείο της Ισπανίας δεν θα πρέπει να επιτρέψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εφαρμόζονται κανόνες που καταστρατηγούν το κοινοτικό δίκαιο. Γιατί αυτός ο κανόνας που έχει αναδρομική ισχύ και προβαίνει σε δίμευση ιδιωτικών περιουσιών, τέτοια χαρακτηριστικά έχει. 14 συνάδελφοι έχουν ζητήσει να μιλήσουν. Έχουμε λιγότερο από 20 λεπτά. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε στην Ελεμέλεια. Ένα λεπτό κάθε βουλευτής. Άλλο χρόνο δεν έχουμε. Χθε ε, ήταν η σειρά μου να μιλήσω και ο κύριος Δέβιτ Λόου δεν ε, μου επέτρεψε να λάβω το λόγο. Έρχομαι από, το Αλικάντε, από τη Σαντα και δεν μου δόθηκε ο λόγος. Κοιτάξτε, χθες είχα τη δικαίωμα να μιλήσετε. Χθες ρώτησα ποιος ήταν παρόν για τις περιφερειακές κυβερνήσει. Έχουμε σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Το Κοινοβούλιο μου δίνει ένα συγκεκριμένο χρόνο. Τώρα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση με του ευρωβουλευτέ. Αν βρεθεί χρόνος, ευχαρίστω θα δώσω το λόγο μετά. Χθε όμω δεν μου δώσετε το λόγο παρόλο που τον είχα ζητήσει. Κολέγκα Μάιερ. Ο κύριος Μέγερ. Θα είμαι λακωνικός κυρία Πρόεδρε. Χθε είπα ότι η πολιτική μου ομάδα δεν είναι κατά του νόμου περί αλλού. αλλά δεν συμφωνούμε με την εφαρμογή του, γιατί διαπιστώθηκαν κάποιες αυθαιρεσίες και ασυμμετρίες στην εφαρμογή του νόμου αυτού. Δεν θα πρέπει εδώ να γίνει συζήτηση ως προς το γενικό συμφέρον ή το γενικό ενδιαφέρον για την ιδιωτική περιουσία. Γιατί αυτή τη συζήτηση την έχει αποφασίσει και το Ισπανικό Σύνταγμα αλλά και ο πρόεδρος Ομπάμα στην Αμερική. Όταν υπάρχουν προβληματικές καταστάσεις ή προβληματικές επιχειρήσεις μπορεί να παρεύει το κράτος και υπάρχει γενικό συμφέρον. Δεν είναι αυτό το ζήτημα όμως. Οι Ισπανικές ακτές είναι από τις ε, πιο ευάλωτες ακτές και τις ακτές που έχουν δεχτεί τις περισσότερες ε, επιθέσεις αστικές στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι χρέος της Ισπανικής κυβέρνησης να προστατεύσει το τοπίο των Ισπανικών ακτών. Διαπιστώνουμε όμως από τις αναφορές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν αυθαίρετη η εφαρμογή του νόμου, ασύμετρη, ιδιότροπη και δεν χρησιμοποιούνται οι ίδια μέτρα και σταθμά για όλους για τα τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα ή για παραδοσιακούς οικισμούς ή για μονοκατοικίες ιδιοκτητών. Δεν εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα στην εφαρμογή του νόμου αυτού. Αυτό καταλάβαμε από τις αναφορές και αυτό είναι και το επίκεντρο της συζήτησης. Η αυθαιρεσία με την οποία εφαρμόζεται μερικές φορές ο νόμος και η ασύμετρη εφαρμογή που διαπιστώσαμε. Πιστεύουμε ότι μερικές φορές αποφασίστηκαν κάποιες ενέργειες χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολιτιστική κληρονομιά. Είχαμε ένα ιστορικό μνημείο εδώ το 1683. Αυτά θα πρέπει φυσικά να διαφυλαχθούν τα μνημεία. Επίσης εφαρμόστηκε, ε, εφαρμόστηκαν δύο μέτρα και δύο σταθμά κατά των απλών ε, πολιτών του Τσοβίτο που κατεδαφίστηκαν τα σπίτια τους ενώ το τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Ρίου Μόλα έχει παραμείνει όρθιο. Δεν πήγαν εκεί οι μπουλντόζες. Οι μπουλντόζες πήγαν σε έναν παραδοσιακό οικισμό ή σε ένα ε, ψαροχώρι απλών ανθρώπων. Εκεί μπήκαν οι μπουλντόζες και κατεδάφισαν τα σπίτια. Υπάρχει λοιπόν ασύμετρη και αυθαίρετη εφαρμογή του νόμου. Θα πρότεινα να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές, να παραμείνουν επιτάπητος και Ελπίζω να επιληθούν τα προβλήματα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να συνεργαστούμε με την Ισπανική Διοίκηση και να επιδιώξουμε ε, διευθέτηση όλων αυτών των προβλημάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρότεινα, κυρία Πρόεδρε, εσείς ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών να στείλετε επιστολή στην Ισπανική Διοίκηση εκφράζοντας το ενδιαφέρον για όλα αυτά τα σημεία και τις αναφορές και να δώσουμε την ευκαιρία στην Ισπανική Διοίκηση να δώσει μια απάντηση, να λάβει μια θέση και εμείς ως Επιτροπή Αναφορών να συνεχίσουμε την περιπτωσιολογική μελέτη όλων αυτών των υποθέσεων. Να παραμείνουν ανοιχτές, παραλαμβάνω, όλες οι αναφορές. Η κυρία Όκεν. Όκεν. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για την εντελεγή παρουσίαση του προβλήματός τους εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω ότι ο νόμος για τις ακτές δεν είναι μόνο εξαιρετικός, είναι και απαραίτητος. Εάν όμως εφαρμόζεται από το εάν είχε εφαρμοστεί από το 1988, τότε ε, θα, είχε, θα είχαν τελείως διαφορετική μορφή οι ισπανικές ακτές. Οποιοδήποτε πηγαίνει στην Ισπανία μπορεί να διαπιστώσει ότι πρόκειται περί καταστροφής και ότι ε, δεν έχει γίνει καμία συντήρηση των ακτών. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι τελείω συμπτωματική εφαρμογή του νόμου. Συμφωνώ με τον κύριο Μαρτίνε, ότι το κοινό συμφέρον ε, θα πρέπει να προηγείται του ιδιωτικού, αλλά ε, ε, αυτό προϋποθέτει ε, σαφείς κανόνες σχετικά με το πώς γίνεται η απαλωτρίωση, ε, προϋποθέτει διαφάνεια και σωστέ διαδικασίες και σωστή ενημέρωση των πολιτών. Αυτό που βλέπουμε σε αυτό το πρόβλημα είναι ότι είναι αυθαιρεσία. Είναι ένας βάλτος όπου οι μεγάλοι μπορούν να προχωρήσουν όπως τους βολεύει, ενώ, ε, ε, ενώ τις επιπτώσεις τις νιώθουν οι μικροί. Γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει να στείλουμε επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση ώστε να φροντίσουμε ε, να, τη, να πληρούνται οι προϋποθέσεις ε, του νόμου, ε, να υπάρχει διαφάνεια ώστε ο νόμος να πετύχει το στόχο του χωρίς να παραβιάζει τα, ε, ε, τα δικαιώματα των ε, πολιτών, διότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν θα πρέπει να παραβιάζεται από την νομοθεσία, ούτε αρκούν απλά οι αποζημιώσεις δεν, νομίζω ότι ακούσαμε πολύ ε, καλές αποδείξεις. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε για πολύ ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Μάιερ. Πιστεύω ότι είναι καλή λύση του προβλήματος. Απ' την άλλη όμως θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν μήπως ε, δεν παραβιάζεται πράγματι ένα κοινοτικό δικαίωμα. Ε, το άρθρο 6 της συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρεται ε, σε δικαιώματα, δεν επιτρέπεται η αναδρομική ισχύς και ε, το δικαίωμα ιδιοκτησίας ρυθμίζεται στην χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε πολλέ περιπτώσεις είδαμε ανθρώπους του οποίους τους ε, κλέβουν το σαλόνι ουσιαστικά όταν επιτρέπεται η χρήση από το κοινό του, ε, της παράκτιας ε, γραμμής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. σύντομη. Προέρχομαι από, την άλλη, από χώρα από την άλλη άκρη της Ευρώπης και εμείς θυσιάσαμε και το λαό μας με εθνικοποιήσεις του 1940 και από εθνικοποίηση πολλών επιχειρήσεων του 1991 και οι διαδικασίε ήταν άδικε έναντι των πολιτών. Η χώρα μου εξέφρασε επιφύλαξη για αυτές τις περιπτώσεις σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από ό,τι ξέρω, για την Ισπανία. Όλες οι περιπτώσεις που ακούσαμε θα μπορούσαν να υποβληθούν και να μελετηθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βέβαια θα χρειαστούν και πολλά λεφτά και πολλής χρόνος και πολλή σκέψη και προσπάθειες. Και σίγουρα στο τέλος η Ισπανική κυβέρνηση, το κράτος μάλλον, θα πληρώσει αποζημίωση διότι σίγουρα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα είναι υπέρ των προσφευγόντων. Γι' αυτό καλώ την Επιτροπή μας να μην προσπαθήσει να λύσει αυτό το πρόβλημα πριν οι περιπτώσεις αυτές έρθουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν τη στρουθοκάμιλο και όταν έχουμε πρόβλημα να χώνουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Πρόβλημα υπάρχει και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο νόμος είναι απαραίτητος, αλλά μερικές φορές έχει κενά και αδυναμίες. Διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες, αποδείχθηκαν από μερικούς. Ακούσαμε ανθρώπινες τραγωδίες στα ισπανικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά. Υπάρχουν αδυναμίες στο νόμο. Δεν μπορούμε να λέμε σε κάποιον που για ένας ολόκληρος είναι ιδιοκτήτης, ε, η οικογένειά του είναι ιδιοκτήτης ενός μήλου και ξαφνικά να χάνει την ε, προσωπική του περιουσία και οι επερχόμενες γενιές ε, να μην μπορέσουν να, να κληρονομήσουν αυτό το αγαθό και απλώς να του δώσουμε 30 χρόνια παραχώρηση. Θα πρέπει η κυβέρνηση να αφήσει έστω και μισάνοιχτη μία πόρτα για να μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματα των αναφερόντων. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις και διεξόδους. Οι αναφέροντες ζήτησαν να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και τώρα θα πρέπει εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Γνωρίζοντας ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι ένα σημαντικό αντιχείο που έχει απήγηση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά μην έχετε και ψευδεστήσεις. Δεν έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή για να τροποποιεί εθνικέ νομοθεσίε. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να παροτρύνουμε την Ισπανική κυβέρνηση, να αφήσουμε ανοιχτέ τι αναφορέ, να στείλουμε επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση ζητώντα πέντε τεινά. Καταρχήν, να επανεξεταστεί ο νόμος περί Αγιαλού, να ακούσει η κυβέρνηση τους θυγωμένους, να ανασταλεί η αναδρομική εφαρμογή του νόμου, να, ανασταλ, να διακοπούν οι οριοθετήσει και επιπλέον ε, να αποφευχθούν οι παρεκτροπές από την εφαρμογή του νόμου. Νομίζω ότι αυτό ζητούν οι περισσότεροι αναφέροντες. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συμπληρώσω αυτά που είπαν συνάδελφοι, ότι Άλλο ένα θέμα είναι η, η ισπανική νομοθεσία, αλλά βλέπω ότι εδώ πέρα υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται να υπάρξει απαλωτρίωση χωρίς αποζημίωση. Δεύτερον, ε, η παραχώρηση χρήσης δεν έχει καμία σχέση με αποζημίωση. Στο σοσιαλισμό τα είδαμε αυτά, ότι ε, γινόντουσαν απαλωτριώσεις αλλά επιτρεπόταν η χρήση της ε, γης. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, συνεχίζει να είναι απαλωτρίωση. Ε, τρίτον, όσον αφορά την, ε, το κτηματολόγιο, αυτά δεν θα πρέπει να μένουν ε, κρυφά από τους ιδιοκτήτες. τρίτον, η αναδρομική ισχύς ενός νόμου. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για απαλωτρίωση. Και το πέμπτο πρόβλημα είναι η αυθαιρεσία πρότασή μου να, ανοίξουμε, να αφήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά. Ως Επιτροπή Αναφορών να στείλουμε επιστολή προς την Ισπανική κυβέρνηση ε, και να τους ε, επιστήσουμε την προσοχή σε αυτά που ακούσαμε σήμερα. Και τρίτον, θα ήθελα η Κομισιόν να κάνει παρόμοια ανακοίνωση προς την ε, Ισπανική κυβέρνηση. Το θέμα δεν είναι ότι ο νόμος δεν είναι αρκετά καλός. Μιλάμε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Κυρία Γκρουνή. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφο Τουρκάη πιο πριν και ο συνάδελφο Γιάρ επίση. Ο νόμος για τις ακτές είναι σημαντικός για να προστατεύει το περιβάλλον, τους διάφορους χώρους και στην Ισπανία καθυστέρησε να ψηφιστεί γιατί οικοδομήθηκαν κτίσματα που άλλαξαν το τοπίο. Εφόσον όμως έγινε σε συμφωνία με ένα ε, ε, σχέδιο χωροταξίας δεν μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε όπως να είναι. Με, με σοκάρισε ιδιαίτερα η προσβολή αυτή του δικαιώματος της ατομικής ιδιοκτησίας Έχουν γίνει οικονομικές επενδύσεις, πρέπει να τη χάνουν συμβασμού. Αν δεν μπορούν να μείνουν τα κτίρια όσοι έχουν, χρειάζεται μια δίκαιη αποζημίωση. Αυτό το δικαίωμα προσωρινής παραχώρησης κονσεσιών απαράδεκτο τελείως. Στη Γαλλία όταν γίνεται απαλωτρίωση, μερικές φορές η αποζημίωση είναι ανώτερη από την τιμή της αγοράς. Μερικοί είναι ικανοποιημένοι όταν τους απαλωτριώνουν την περιουσία τους. Χρειάζεται δράση, δεν πρέπει να κλείσει η αναφορά αυτή. Πρέπει να την παρακολουθήσουμε από κοντά, από εδώ και μπρος, για να πάρουμε απαντήσεις. Μπορεί να τίθεται κάποιο θέμα σχέση με το κοινοτικό δίκαιο, αλλά εμείς ως Επιτροπή Αναφορών που πρέπει να εισακούμε τους πολίτες πρέπει να είμαι ευαίσθητοι στον αριθμό των αναφερόντων καταρχήν που μας μίλησαν σήμερα και πολλών άλλων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άντερσεν. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι περιπτώσεις που ακούσαμε σήμερα αφορούν το δίκαιο της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά αποκαλύπτουν και την κατάσταση χάους με τον οποίο ε, ασκείται η χωροταξιακή πολυδομία στην Ισπανία. Είναι περίεργο το ότι η Ισπανική κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει του πολίτε. Η Ισπανική οικονομία περνάει σοβαρή κρίση που ξεκίνησε μέσω των ακινήτων και των κατασκευών. Όλοι υπέφεραν από την κυριοδοσκοπία και από την εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου για τον Αγιαλό και άλλων οικιστικών νόμων. Καλό θα ήταν να γίνει μια συζήτηση να μην πηγαίνουν επιδοτήσεις στην Ολομέλεια, να μην πηγαίνουν επιδοτήσεις στις περιοχές αυτές. Το προσπάθησα, προσπάθησα να με υποστηρίξουν άλλε ομάδε. Τρει εκθέσει πέρυσι από την Ομέλεια, κανένα αποτέλεσμα. Ήρθε η στιγμή να επιβάλλουμε δια τη βίας να πετύχουμε βία, δηλαδή να μπλοκάρουμε τις επιδοτήσεις προς την Ισπανδία. Η περίπτωση τη Ισπανία δεν είναι και πολύ διαφορετική από την Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Νίκολσον. Ευχαριστώ. Ήρθα εδώ σήμερα γιατί μου το ζήτησαν οι εκλογείς μου. Έχω μπουχτίσει από τους εκλογείς μου κάθε εβδομάδα 10 με 20 άτομα έρχονται και καταγγέλνουν ότι χάσαν τα λεφτά τους όχι μόνο από την Ισπανία και άλλες χώρες. Βουλγαρία, για την, Τουρκία, ισχύει. Και είμαι πολύ απογοητευμένος ή έχω διαβάσει επιστολές ως Ευρωβουλευτής. Έχω γράψει τη μόνιμη Ισπανική αντιπροσωπεία στι Βρυξέλλε. Έχω γράψει στον Ισπανό Πρωθυπουργό, στι περιφερειακέ αρχέ. Ούτε καν απάντηση δεν πήρα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον Είχαμε μια πολύ καλή παρουσίαση, δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που ακούσαμε. Τι θα γίνει από εδώ και μπρό. όσο μας αφορά. Αν το αφήσουμε θα περάσει και σε άλλες χώρες. Η Τουρκία θέλει να ενταχθεί. Πριν ενταχθεί θα πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Να σταλεί μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και τις Ισπανικές Αρχές αλλά αν κρίνουμε από το παρελθόν δεν νομίζω θα είναι αποτελεσματικό. Να γράψουμε μια επιστολή, αλλά να επιφυλαχθούμε και για επιπλέον μέτρα, διότι αξίζει για τον κόσμο αυτό αυτή η προσοχή. Σαλαβράκος. Ε, κύριε Πρόεδρε ε, και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι κανένας μας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση, κανένας μας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση αυτών των ανθρώπων που ήρθαν σήμερα εδώ να μας αναπτύξουν το πρόβλημά τους. Βέβαια, εν ονόματι των μεγάλων ιδεών πάντοτε γίνονται και τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Και η δημόσια ωφέλεια που είναι μια μεγάλη ιδέα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά. Και όταν μιλάμε σωστά πρέπει εάν θέλουμε να απαλωτριώσουμε ιδιοκτησίες να υπάρχει πλήρης αποζημίωση, δηλαδή τόση ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση της περιουσίας με κάποια ίσης αξίας άλλη περιουσία. Από ό,τι κατάλαβα δεν συμβαίνει αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Ε, βεβαίως δεν μπορούμε νομικά να μπούμε λόγω της αρχής της επικουρικότητας στις εσωτερικές διατάξεις ενός άλλου κράτους. Η εφαρμογή όμως του νόμου αυτού είναι προφανώς ότι είναι στρεβλή και προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των αναφερόντων και κατά την πείρα μου οφείλεται στην, και δημιουργεί ε, ε, κακό στα δικαιώματα των μικροϊδιοκτητών ενώ δεν πλήττει τους μεγάλους εξυπηρετώντας μια αυθαιρεσία. Λοιπόν θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με την άποψη του κ. Μάγερ να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να κάνουμε τα δέοντα προς την Ισπανική κυβέρνηση. Er Καταρχήν να πω ότι μιλάμε για παραδόσεις σε κράτη-μέλη, οι οποίες είναι διαφορετικής φύσης και εδώ πέρα έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα. όταν ε, αγοράζει κανεί σε σπίτι, ουσιαστικά αγοράζει κομμάτι του, της πολιτιστικής παράδοσης σε ενός ε, κράτους. Ε, υπάρχουν δηλαδή περιορισμοί στο κατά πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους αναφέροντες. Αλλά βλέπουμε εδώ πολλά σημάδια αυθαίρετης εφαρμογής του νόμου. Και ε, πέρα από την πρόταση του κυρίου Μάγερ θα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Θα ήθελα από την Κομισιόν σαφή απάντηση ε, που έχουν χρησιμοποιηθεί οι ε, πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προγράμματα αυτά. Εάν δεν μπορούμε άμεσα να επέμβουμε λόγω της επικουρικότητας, θα πρέπει να φροντίσουμε τουλάχιστον που, ε, μπορούν, που μπορεί να σταματήσει η χρηματοδότηση για τέτοια ε, έργα. Και να δούμε έμεσα πού δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεσμεύεται και το ευρωπαϊκό και το τοπικό επίπεδο από αυτά. Και επίσης όσον αφορά αυτά που ακούσαμε. Κύρια Πρόεδρε, στο δικό μου Δήμο είδα είδα ότι όταν ε, κάποια ε, χρήματα δίδονται σε, σε κάποιες οικογένειες για, για δημογραφικούς λόγους, ε, παρεμβαίνει η Επιτροπή. Αλλά εδώ πέρα όταν, όταν έχουμε μεγάλο κράτος μέρος, έχουμε την εντύπωση ότι κανένας δεν παρεμβαίνει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στην ε, αναφορά αυτή. Ευχαριστώ. Κύριος Μαρτίνες. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με μεγάλη ηρεμία, αλλά να είστε συγκαταβατικός και να είστε και επίοικείς με μένα και με το χρόνο μου, γιατί ήμουν ο μόνος που δέχτηκε προσωπικές επιθέσεις και υπενιγμούς. Θα ήθελα καταρχήν για να διευκρινίσω τα πράγματα να πω ότι σέβομαι όλους τους αναφέροντες και θα ήθελα να πω σε ορισμένους από αυτούς ότι εγώ προσωπικά πλήρωσα με χρόνια φυλακής και μερικά νύχια από δάχτυλα το δικαίωμα στην ελευθερία, το δικό μου και το δικό σας και έκανα χρόνια ολόκληρα προσπάθειες για να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη μορφή που έχει σήμερα. Όχι όπως κάποιοι συνάδελφοι που στο πρόγραμμα και στις δράσεις τους φέρουν ως στόχο την εξαφάνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αν εξαφανιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αν είχε εξαφανιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχατε σήμερα αυτό το δικαίωμα να έρθετε εδώ και να ασκείτε το δικαίωμά σας ε, ε να εκφέρετε ελεύθερα τη γνώμη σας και να υποβάλλετε τις αναφορές σας. Θα ήθελα να πω σε όλους ότι ευτυχώς αυτός που προσδιορίζει τι είναι συνταγματικό στην Ισπανία και τι όχι, δεν είναι μια ομάδα πολιτών, δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το συνταγματικό δικαστήριο της Ισπανίας. Το συνταγματικό δικαστήριο της Ισπανίας χαρακτηρίζει συνταγματικό ή αντισυνταγματικό ένα νόμο. Μπορεί η αποφάσεις του να να μην μα βρίσκει σύμφωνο. Μπορεί ένα νόμο να μα αρέσει και άλλος όχι, αλλά αυτό ο αρμόδιο να αποφασίσει είναι το συνταγματικό δικαστήριο. Και η παραχώρηση χρήση είναι ένα τρόπο αποζημιώση. Αυτό το έχει κρίνει ω θεμητό τρόπο αποζημίωση το ίδιο το συνταγματικό δικαστήριο τη Ισπανία, που είναι αρμόδιο, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτή την απόφαση. Δεν είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρίνει κάτι τέτοιο. Όντως, ο νόμος περί και ακτών είναι πολύ περίπλοκος και η εφαρμογή του είναι περίπλοκη. Γι' αυτό και υπήρξαν αρκετές διαμαρτυρίες. Πάντως είναι πολύ προοδευτικός, από τους πιο προοδευτικούς νόμους ε, για τις ακτές και εμείς θα παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη της υπόθεσης και φυσικά θα ακούσουμε τους ε, και θα κρίνουμε περιπτωσιολογικά, θα αξιολογήσουμε περιπτωσιολογικά κάθε αιτίαση. Και η προηγούμενη κυβέρνηση ε, που ήταν από άλλη παράταξη εφάρμοσε τον νόμο και δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση και μάλιστα οριοθέτησε πολύ περισσότερα χιλιόμετρα η προηγούμενη κυβέρνηση από ότι η τωρινή κυβέρνηση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους αναφέροντες που έδειξαν εμπιστοσύνη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι οι εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών είναι γνωστές και περιορισμένες. Δεν μπορούμε να έχουμε αρμοδιότητε περισσότερε από ό,τι έχουμε. Δεν θα πρέπει να έχουν ψευδεστήσει ή να πλανώνται μερικοί ε, ότι έχουμε περισσότερε αρμοδιότητε από αυτέ που έχουμε πραγματικά. Ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα αναφέρω ούτε αυτή την κυβέρνηση, ούτε προηγούμενες κυβερνήσεις της Ισπανίας, γιατί και έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι η σημερινή κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από την κατάσταση στο παρελθόν. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα, ακούσαμε ε, αισθήματα, συναισθήματα και μερικές φορές είδαμε και κάποια δάκρυα εκνευρισμού, ματέωσης, απογοήτευσης, ανημποριάς. ακούσαμε περιπτώσεις ε, της τη της Μπράβα, τη Ανταλουσία. Είδαμε ότι είναι αναδρομική παράνομη εφαρμογή του νόμου, εφαρμόζεται αυθαίρετα και παραβιάζει θεμελιώδη δικαίωμα όπω είναι αυτό τη ατομική ιδιοκτησία. Επίσης υπήρξε μία ομόφωνη αίτηση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει κάτι και να προσφύγει στο δικαστήριο. Ε, δεν θα πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, να μην μείνουμε απαθείς από αυτά, σε αυτά που συμβαίνουν στην Πάλμα, στη Φορτεβεντούρα, στο Τσοβίτο και σε πολλοί άριθμα άλλα μέρη. Το η... Ισπανική κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου, να προστατεύσει το... την ατομική ιδιοκτησία, να προστατεύσει τα δικαιώματα κυριότητα και να σταματήσει τι ε, αυθαίρετε καταδαφίσει. Σε αυτή την προσπάθεια θα υποστηρίξουμε του ε, αναφέροντε. La η κυρία Σταρίας. Οι νομοθέτες στα διάφορα κοινοβούλια, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν αρμοδιότητα την κατάρτιση νόμων. Και η εκτελεστική εξουσία, οι κυβερνώντες, έχουν την αρμοδιότητα της εκτέλεσης εφαρμογής του νόμου, εφαρμόζοντας όμως και την κοινή λογική. Θα πρέπει οι κυβερνώντες να δουν αν είναι λειτουργικός ένας νόμος, αν επιδέχεται βελτιώσεις ή όχι. αν Έχουμε περίπτωση νόμου που, όπως στο νόμο περιακτών, μετά από 20 χρόνια εφαρμογής διαπιστώνουμε ότι εφαρμόστηκε αυθαίρετα και άδικα, ο σωστό κυβερνών θα πρέπει να ανασκουμποθεί και είτε να αναθεωρήσει τον ίδιο τον νόμο, είτε να αναθεωρήσει την εφαρμογή του σε περίπτωση που η εφαρμογή αυτή οδήγησε σε αδικίες. Απευθύνω έκκληση προς την Ισπανική κυβέρνηση να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Γιατί ήδη το 2006 ο πρόεδρο Απατέρο, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ε, υποσχέθηκε μία δίκαιη οριοθέτηση για το νησί της Φορμεντέρα και η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κυρία Βέγα. Και είδατε τις τεράστιες ασδικίες που είχαμε, γιατί μένουν άθικτα τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα στις παραλίες, ενώ μικρά κτίσματα και ε, ιδιωτικές ε, οικίες ε, κατεδαφίζονται. Θέλουμε μια δίκαιη οριοθέτηση για τη Φορμεντέρα και ζητούμε από την κυβέρνηση Ισπανίας και από τον κύριο Σαπατέρο να τηρήσει τις υποσχέσεις που έδειξε, να τηρήσει το λόγο της. Η κυρία Χιμένες. Χθες και σήμερα ακούσαμε τα ίδια λόγια σε πολλές γλώσσες. Αυθαιρεσία, παραπληροφόρηση, κατάχρηση ε, σε ό,τι αφορά τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, άδικες απαλωτριώσεις, χωρίς δίκαιες αποζημιώσεις. Δύο μέρες ακούσαμε τις ίδιες καταχρήσεις σε πολλές γλώσσες. Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν, γιατί ζητήσαμε να μείνουν ανοιχτέ αυτές οι αναφορές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αρχιοθετηθούν και θα ήθελα να πω σε όλα τα θύματα, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι θύματα όλοι αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό ήρθαν σήμερα να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους. Για, για είναι πολύ εύκολο να μιλάμε ε, δημοσίω, αλλά για τους ανθρώπους αυτούς είναι πολύ δύσκολο να έρχονται και να εκφωνούν μια ομιλία μπροστά σε ακροατήριο. Και φυσικά υπάρχει συγκινησιακή φόρτιση, γι' αυτό και θα πρέπει να του εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια που αξίζουν. Σα υπόσχομαι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα αιτήματά σα. Ευχαριστώ κυρία Να μην προσθέσω κι εγώ σε όσα ακούσαμε. Απλώς καταθέτω κι εγώ τη φωνή μου. Οι αναφορές πρέπει να μείνουν στο τραπέζι ανοιχτές και πρέπει να γράψουμε και στην Ισπανική κυβέρνηση. Ο κύριος Αρίας. Θα είμαι κι εγώ τηλεγραφικό, γιατί ελάχιστο χρόνο μας δώσατε, όπως και στου υπόλοιπου. Έχω σοβαρέ αμφιβολίες για τον νόμο, το είπα και χθε το επαναλαμβάνω και σήμερα. Έχω αμφιβολίε αν είναι ένας καλός νόμος που ισχύει πάνω από 22 χρόνια και μπορεί να είναι θεωρητικά καλός για να προστατεύσει την ισπανική ακτογραμμή, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι καλός για να προστατεύει τα δικαιώματα ατομικής ιδιοκτησίας ε, των πολιτών ε, που έχουν περιουσία στις ευρωπαϊκές ακτές. Φαίνεται ότι θυγόμενοι είναι πάνω από 300.000. Δεν νομίζω ότι είναι, ε, επιδέχονται ερμηνείε, διαφορετικές οι νόμοι. Βέβαια, κανένας νόμος δεν είναι τέλειος, οπότε αν διαπιστώνονται αδυναμίες, καλό είναι να αναθεωρούνται αυτοί οι νόμοι. Ήρθε η στιγμή για τη μεταρρύθμιση και δεδομένου ότι η εφαρμογή του νόμου αυτού δημιούργησε πρόβλημα, θα πρέπει επιτέλου ο νόμο περιακτών να αναθεωρηθεί. Πιστεύω ότι υπάρχουν και συγκαλυμμένα, κρυφά ελαττώματα στο νόμο και αυτά τα ελαττώματα άρχισαν πια να βγαίνουν στην επιφάνεια. Και ένα λεπτό έχετε κι εσείς το λόγο από την τοπική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να επαναλάβω όλα αυτά τα θέματα που αναφέρθηκαν. Το μόνο που θα ήθελα να πω ότι οι μικρές τοπικές διοικήσεις βρίσκονται τελείως ανήμπορες απέναντι στην εφαρμογή του νόμου αυτού. Και όταν οι οριοθετήσεις γίνονται σε ε, βιομηχανίες ή μικρά μαγαζάκια που αποτελούν τη βάση της οικονομίας μικρών δήμων και κοινοτήτων και η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται ότι όταν εφαρμόσει τις οριοθετήσεις, τις απαλωτριώσεις και τις παραχωρήσεις θα διακυβεύσει την επιβίωση μικρών τέτοιων επιχειρήσεων που είναι οι επιχειρήσεις που ε, δημιουργούν ζωή σε πολλές περιοχές όπως είναι το πάρκο της Αλικής ε, του Σανταπόλα που είναι μια τη η αλική που, χρησιμοποιεί, που κατασκευάστηκε για την εξόρυξη άλακτος, αν διακυβεύσουμε τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες, πώς θα μπορέσουμε να ε, κρατήσουμε ζωντανή την αλική, γιατί αν εφαρμόσετε την οριοθέτηση, θα αποξηρανθεί η αλική και η περιοχή μου θα χάσει μια, ένα πολύ σημαντικό αξιοθέατο που προσελκύει τον τουρισμό κύριε Πρόεδρε. είμαι πάρα πολύ σύντομο. Όλοι συμφωνούμε ότι, και μια περί... ότι πρόκειται για μια περίπτωση πάρα πολύ σύνθετη και αυτό οφείλεται στην χαρακτήρα, στο γεωγραφικό χαρακτήρα των ακτών της Ισπανίας. Δεύτερον, είναι θέμα των επικυρίαρχων δικαιωμάτων μιας χώρας να νομοθετεί μέσα στα πλαίσια της επικουρικότητας. Τρίτον, δεν συμφωνώ και δεν θα συμφωνήσω ποτέ να παίξουμε πολιτικά με το θέμα αυτό. Μερικοί το παίζουν αθώοι, ξέροντας ότι στην Ισπανία από την έγκριση του νόμου και μετά υπήρξαν διαδοχικές κυβερνήσεις του Λαϊκού και του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Τέτατο, συμφωνώ ότι παρά την θεσμική περιπλοκότητα του θέματος που οφείλεται σε έναν βαθμό στην ε, ιστορική οργάνωση και παράδοση του Ισπανικού κράτους υπάρχει μια διαχείριση στο πώς εφαρμόζεται ο νόμος αυτός και ποιες είναι οι επιπτώσεις του και χρειάζεται μια, μια ανακολουθία στη δράση αυτή. Ελπίζω η Ισπανική κυβέρνηση, τον οποίων εκπρόσωποι παρίστανται φαντάζομαι, να μας πληροφορεί περιοδικά για το πώς ε, προσαρμόζει και εφαρμόζει αυτό το νόμο. και δεν δέχουμε τη σύνδεση με την Ισπανία, με χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης ή να σταματήσει η χρηματοδότηση της Ισπανίας από την Ένωση. Γιατί η φιλοσοφία πίσω από τα ταμεία αυτά και τα κονδύλια αυτά είναι εντελώ διαφορετική. Πρόεδρος. Τελευταία παρέμβαση, παρακαλώ. Τελευταία παρέμβαση, συναδέλφου. Τελευταία παρέμβαση. Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή την πορεία της έκθεσης Άουγεν και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι χθες ήρθε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης και άκουσε πολλές παρατηρήσεις, κάτι που δεν συνέβαινε προηγούμενες κυβερνήσεις για πολύ σημαντικές υποθέσεις που είχαμε επεξεργαστεί. Δεν είχαμε τότε εκπροσώπους προηγούμενης κυβέρνησης. Τουλάχιστον η Ισπανική κυβέρνηση έστειλε έναν εκπρόσωπο στην περίπτωση αυτή για να ακούσει τα παράπονα των αναφέροντων. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η χειρονομία της Ισπανικής κυβέρνησης που ήρθε εδώ και άκουσε τις αιτιάσεις των ετούντων. Επίσης θα ήθελα, συνάδελφοι, εσείς που ακούσατε στον τύπο ή διαβάσατε στον τύπο στις χώρες σας ότι δεν ξέρουν οι αλλοδαποί που αγόρασαν στην Ισπανία τι γίνεται με την εφαρμογή αυτού του νόμου. Ο νόμος αυτός είναι, είναι και σέβεται και το κοινωτικό κεκτημένο. Το σημαντικότερο είναι να ακούσουμε τα παράπονα των αναφερόντων, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και να βρούμε κάποιες λύσεις και με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις αλλά και με την κεντρική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Η πλειοψηφία των συναδέλφων λοιπόν είναι υπέρ του να παραμείνει ανοιχτό το θέμα αυτών των αναφορών. η Ισπανική κυβέρνηση να γράψει μια επιστολή. Νομίζω η πλειοψηφία αυτό ζήτησε. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ πολύ, θα σας ζητήσω να ψηφίζουμε. Έχουμε έναν αναφέροντα που μας περιμένει από χθε. Έχω την υποχρέωση να του δώσω το λόγο. Άρα να περάσουμε στην επόμενη αναφορά. Νομίζω όλοι μιλήσαμε, εξαντλήσαμε όλο το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας ο καθένας. Θα απευθυνθούμε στην κυβέρνηση διότι η απόλυτη πλειοψηφία των συναδέρφων ζήτησε να γράψουν μια επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση να ζητήσουμε διευκρινήσει για όλα τα σημεία που ανεφίησαν στη συζήτηση χθε και σήμερα και να ζητήσουμε και από την Κομισιόν να απαντήσει συγκεκριμένα στο ερώτημα της υποτιθέμενης παραβίασης που ετέθη άρθρα της συνθήκης Σύμβαση Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα γράψουμε δύο επιστολές για διευκρινήσεις. Και θα ξαναπιάσουμε τη συζήτηση αργότερα. Η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει λεπτομεριακά στο σημείο με αυτό. Για το τι συζητήθηκε εδώ. Κλείνω με την αναφορά αυτή και περνάμε στην αναφορά υπαριθμό 18. do la parola al petente James Lanney. Vi prego di uscire in silenzio perché abbiamo solo... James Lanney, 18. Παρακαλώ, έχουμε 5 λεπτά μόνο για τον αναφέροντα που έχει το δικαίωμα με όλους σας.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 Παρακαλώ, λέγομαι James Loney, είμαι ο αναφέρον και με τη ομάδα δράση του Nevit Lask στην Ιρλανδία. Μια σύντομη εισαγωγή στα Ιταλικά προς την πρόεδρο την κυρία Ματσόνη, η οποία όμως έχει φύγει. Αγαπητή κυρία Ματσόνη, έχετε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη γιατί ότι δώσατε στο Action Group του Nevit Lask στην ομάδα δράσης την ευκαιρία να απευθυνθούμε στην Επιτροπή Αναφορών για να σας παρουσιάσουμε και να συζητήσετε τον προβληματισμό μας σχετικά με την πρόταση σχετικά με την υπερχοματερή στην ε, κοινότητά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μάλλον δεν γνωρίζετε την υπόθεσή μας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον συνάδελφο Ντέκλαν, ο οποίος είναι μηχανικός και ότι θα παρουσιάσει την περίπτωση αυτή. Uh, Fingal County Council is proposing to put... Το Φίνγκαλ ε, ε, ε, το, τοπική αυτοδιοίκηση ε, προτείνει να εγκαθίσει μια από τι πιο καθαρέ χωματερέ στην Ευρώπη. Αυτό όμω παραβιάζει ε, την οδηγία για τι χωματερέ, την οδηγία για το πλαίσιο για το νερό, για τα υπόγεια ύδατα, την οδηγία για τι χωματερέ, την οδηγία ΑΕΑ και ε, και την οδηγία για την στρατηγική για το περιβάλλον γιατί υπάρχει κίνδυνος για υπόγεια είδα, τα μακροπρόθεσμα και για την ατμόσφαιρα. Βέβαια, Ο χάρτης αυτός σας δείχνει πώς είναι οι υπόγειες πηγές στην Ιρλανδία. Έχουμε ένα υπόγειο υδροφορίζοντα, Fisher Bedrock, όπως λέμε στο Fingal, με δυναμικό περίπου 40 εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα. Η ομάδα μας ε, όρισε ε, την, γεωλογικό survey της ε, Ιρλανδίας να μας δώσει έναν χάρτη δάτων της περιοχής. 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στο Φίγγαν συγκεκριμένα 450. Απασχολούνται 20.000 άτομα στην περιοχή με παραγωγή φυτικού προϊόντος με ένα καθαρή παροχή νερού. Η κοινότητα μας είναι 206 άτομα και η η παραγωγή αυτή είναι η κύρια απασχόληση και είναι γνωστό ως ε, από τα κύρια κέντρα παραγωγής αυτού του προϊόντος στην Ιρλανδία. 55% των επόμενων προϊόντων παράγονται από την δική μας κοινότητα. Εξαρτώμαστε από το καθερό και επαρκές είδωρ, από τον υδροφόρο αυτό ορίζοντα για ίδρυυση και κατεργασία του προϊόντος. Βέβαια, ο κλάδος αυτός ε, δεν έχει ε, παρακολουθηθεί ως μέρος του AEI. Μόνο μια έρευνα ε, των, ε, φρεάτων έγινε από την RPS. Αυτή η χωματερή θα οδηγήσει 26 άτομα να χρειαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους και από τη γη τους. 210 εκτάρια πολύ καλής γεωργικής γης θα καταστραφούν για πάντα. Το όνομα Νέβιτ προέρχεται από την κελτική λέξη Νέμετον, που σημαίνει ιερό. Το Νέβετ είναι το μόνο, ο μόνος επιζών χώρο στην Ευρώπη με αυτό το όνομα. Οι Ιρλανδικές αρχές δεν έκαναν μελέτες αρχαιολογικές στο χώρο. Αυτό είναι μια απόφαση μεροληπτική υπέρ της χωματερής. Η κοινότητά μας στο δημοτικό σχολείο είναι σε απόσταση 500 μέτρα από τη χωματερή και έχει δοθεί έγκριση για ένα νέο σχολείο 300 μέτρα από τα όρια της χωματερής. Η AES λέει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά λόγω σκόνης, ε, αναθυμιάσεων ή αερίων που θα βγαίνουν από τη χωματερή αυτή. Η εμπειρία είναι τελείως διαφορετική σε άλλα της Ιρλανδίας. Δυστυχώς η χωματερή είναι σημαντική πηγή εισοδήματος και η αρχή ο Ριπέρον πληρώνει χρησιμοποιείται εδώ. Η Ιρλανδία ε, έχει δώσει την άδεια για το διπλάσιο στην έκθεση αυτής της ε, χωματερίας. Δόθηκε έγκριση να υπάρχουν δύο πορτεφροτήρες 15 χιλιόμετρα βόρεια στον χώρο και ένα 25 χιλιόμετρα στον νότο με συνολική απόδοση 800 εκατομμύρια κιλά το χρόνο. Επιπλέον θα χρησιμοποιείται και για το Δουβλίνο με δυναμικό 350 εκατομμύρια κιλό το χρόνο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της, ε, ε, το ότι υπάρχουν πάρα πολλές χωματερές και συγχρόνως μειώνεται το κόστος όταν χρησιμοποιείται η χωματερή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος υποστηρίζει αυτό, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση μένει στις παλιές ιδέες και στο τι θα κερδίσουν. Το να έχουμε καθαρό νερό είναι ακρογωνίας λίθος για μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Στην Ελλάδα εξαρτώμαστε και από τα επιφανειακά ύδατα για τη βιομηχανία. 16% μόνο προέρχεται από υπόγειες πηγές. Γι' αυτό το επίγειο είδωρ, επειδή θα ρηπανθεί από, σε περιπτώσεις πλημμύρας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας. Το περιβάλλον της Ιρλανδίας απειλείται σοβαρά από τις εσφαλμένες πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα ε, υδάτινων πηγών και διαχείρισης των αποβλήτων. Ο επόμενο ομιλητή θα σα αναφέρει τι διάφορε παραβιάσει οι οποίε έγιναν στον τομέα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ο, η χωματερή που προτείνεται στον ΕΒΙΤ με χωρητικό 400.000 τόνους είναι, αποτελεί ένα στοιχείο για το ε, σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για